Hello. Good afternoon to everybody. Γεια σας, καλησπέρα. Ας ξεκινήσουμε. Οπότε. Έχετε λάβει όλη την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις, αυτή εγκρίνεται. Περνάμε στο δεύτερο σημείο ανακοινώσεις της Προέδρου. Οπότε τώρα πρέπει να διαβάσω εδώ πέρα τα διάφορα. Λοιπόν, η Επιτροπή μας έλαβε τρία σχέδια διορθωτικού στην θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που εγκρίθηκε στην πρώτη ανάγνωση στις 16 Απριλίου. Πρώτος ο κανονισμός ε, που αλλάζει τους κανονισμούς ε, EBA, κανονισμός ε, ΕΙΟΠΑ 2010, ε, ΕΣΜΑ 1095-2010. ΜΥΦΙΡ, ο κανονισμός 600 κάθετος του 2014, benchmarks, ο κανονισμός του 2016-1011, επίσης transfer funds, μεταφορά πόρων, ο 807 του 2015 και κατόπιν έχουμε την οδηγία που τροποποιεί τις ε, ε, εξής οδηγίες, MIFID 2 του 2014 κάθετος 65 ΕΕ κατόπιν η οδηγία για το αξιόχρονο υπαριθμό 2, οδηγία 2009 κάθετος 138 και η EMLD, η οδηγία του 2015 κάθετος 849 και τέλος έχουμε τον κανονισμό ο οποίος τροποποιεί τον κανονισμό ECRB η διαδικασία του 2017 με 232 και τα σχέδια κείμενων όλα έχουν διαβαστεί στα μέλη τη Επιτροπής ε, Οικονομικών Υποθέσεων την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου σε όλε τις γλωσσικές εκδοχέ με τον ε, με τη διάταξη 241 του κανονισμού μα, εάν δεν υπάρχει κάποια ένσταση από την Επιτροπή, τότε πρόκειται αυτά τα διορθωτικά να υποβληθούν στο Κοινοβούλιο και αυτά πρόκειται να ανακοινωθούν στην πρώτη ολομέλεια του νευρίου και θα θεωρηθούν εγκεκριμένα εκτό εάν ε, ε, μια πολιτική ομάδα ε, ή μέλη που φτάνουν μέχρι το 138 ζητήσουν να γίνει ψηφοφορία. Τώρα, έχουμε τα σχετικά με τους τριμερείς διαλόγους που άρχισαν την περασμένη εβδομάδα, δηλαδή πριν από δύο εβδομάδες. Οπότε έχουμε ε, τους ε, φακέλους για το crowdfunding, ο τριμερείς διάλογος 22-19, καλούμε τις απόφασεις μας να αρχίσουν δύο οργανικές διαπραγματεύσεις μετά την δεύτερη ανάγνωση στις 20 Σεπτεμβρίου, πρώτο διερευνητικό τμήμα διάλογο είναι στι 22 στο Στασβούργο και το Κοινοβούλιο αλλά και το Συμβούλιο παρουσίασαν τι τοποθετήσει του και ο πρώτο τμήμα διάλογο τόνισε ότι υπάρχουν σημαντικέ διαφορέ μεταξύ των ΜΕΝ και των ΔΕ και συγκεκριμένα ο βαθμό εναρμόνιση του ευρωπαϊκού καθεστώτο για τι υπηρεσίε crowdfunding και του παρόγου αυτών και το πεδίο εφαρμογή αυτή τη πρόταση θα είναι σημαντικό θέμα ζήτηση στον επόμενο τριμερή διάλογο που είναι στι 6 ενδεκάτου. Ε, Άλλο τριμερή διάλογο που αφορά τι ε, βιώσιμε επενδύσει τη 23η δεκάτου του 19 κατόπιν τη έγκριση σε μια κοινή συνεδρίαση τη ΕΚΟΝ και τη ΕΝΒΙ όσον αφορά την απόφαση να αρχίσουν οι διαπραγματεύσει τη Δευτέρα 21 δεκάτου το Συμβούλιο παρουσίασε τα βασικά στοιχεία της γενικής προσέγγισης όπως συμφωνήθηκαν από την Κορεπέρ στις 25 Ενάτου. Παρουσίασε το Κοινοβούλιο τα βασικά στοιχεία της θέσης του που συμφωνήθηκαν στην πρώτη ανάγνωση κατόπιν των εισηγήσεων και την πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκλήθη να προσφέρει πλέον πληροφορίες τη σχέση μεταξύ της πρότασης ταξόνομη και ε, του πρόσφατου κανονισμού σε σχέση με τις αποκαλύψεις, το disclosure και τα δύο μέρη συμφώνησαν να υπάρξουν τριμερείς διάλογες στις 20 και 27 ενδεκάτου αλλά και 3 12 του επόμενη ανακοίνωσή μου αφορά μια περίληψη των αποφάσεων των συντονιστών ε, στις 11 ενδεκάτου και στη συνέχεια στις 16 ενάτου και 2 δεκάτου. Πρώτα πρώτα όσον αφορά το πλαίσιο διακυβέρνησης για το ε, δημοσιονομικό όργανο σύγκλησης και την αγωνιστικότητας για την Ευρωζώνη και επίσης την απαλλαγή ε, της ESA ε, που αφορά το Προεδρείο. Και συμφωνήθηκε και αυτό εκκρεμεί ακόμα ότι θα πρέπει να γίνουν να ε, σχετική προθεσμία για τις ε, τροπολογίες και συμφωνήθηκε ότι αυτές που υποβλήθηκαν την 8η θητεία ε, έχουν λήξει και τώρα θα πρέπει να δούνε τι θα κάνουν οι πολιτικές ομάδες και αυτό αφορά το δημοσιονομικό σύμφωνο αλλά επίσης και το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων όπως και την σταθεροποίηση των ευρωπαϊκών επενδύσεων και είπαμε ότι και εδώ θα πρέπει να συνεχίσουν να ισχύουν αυτοί που έχουν οριστεί ως συγκητής και σκιώδεις συγκητές. Ε, βέβαια όχι αυτοί που τώρα δεν είναι πλέον βουλευτές. Επίση, είπαμε ότι συμφωνούμε για τα ερωτηματολόγια για την κυρία Βεστάγκερ, τον Πρόφσκης και Τζεντιλόνη, να συνεχίσουμε τη συνεργασία με την ομάδα εργασία για την Τραπεζική Ένωση, ε, για την ομάδα εργασία του ανταγωνισμού, όπως επίσης και χρηματοδοτική ε, ε, αρρωγή και να συγκροτηθούν καινούργιε ομάδες εργασίας για τις χώρες υποψήφιες για την Ευρωζώνη και FinTech. Και είπαμε ότι πρόκειται να συγκροτηθεί επίσης μια υποεπιτροπή για θέματα φορολογικά, υποεπιτροπή της ΕΚΟΝ. Πέμπτη ανακοίνωση. Το κυκλικά εναλλασσόμενο πρόγραμμα της Επιτροπής είπαμε ότι θα γίνουν εξή προτάσεις ενημερώσεων, πράσινη οικονομία, ε, κάτι δέν ε, νομίσματα, fintech και τεχνητή ευφυΐα, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες ε, αξιολόγηση, συγγνώμη, φορεί αξιολόγηση, νομισματική πολιτική, νομισματική ένωση, τροπική ένωση και καταπολέμηση πλησίματο χρημάτων, του ξεπλήματο χρημάτων. Και είπαμε ότι οι προτάσει πρόκειται να υποβληθούν στου νομιστές για έγκριση τον ε, διορισμή. Ευρωπαϊκή Στατιστική Συμβουλευτική Επιτροπή ζητήθηκε από τις ομάδες να αποσταλούν γραπτές προτάσεις για να οριστεί εμπειρογνώμονας από το Κοινοβούλιο. Έβδομο, εξέταση πράξεων κατεξουσιοδότηση και εφαρμοστικών μέτρων εγκρίθηκαν οι νέες κατευθυντήριες γραμμές ε, και αποφασίσαμε να οργανώσουμε μια συνεδρίαση για να εξετάσουμε τα θέματα αυτά. 8 δημόσια ακροάση μέχρι τον Ιούνιο του 2020. Δεν έχει ζητηθεί κάτι αυτή τη στιγμή. Ένα το αποστολές το 2020 συμφωνήσαμε σε εξής αποστολές. Πρώτον, αποστολή στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, Στρασβούργο Δευτέρα το πρώτο τρίμηνο, Βασιλεία, Στρασβούργο Δευτέρα Άνοιξη του 2020, 12 βουλευτές, ε, Παρίσι, ΟΣΑ και Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, 6 και 7 Απριλίου, 7 ε, βουλευτές, Σύνη Πρόεδρος, Βερολίνο, 18-19 Μαΐου 6 βουλευτές, Ουάσιγκτον, 20-23 Ιουλίου 7 βουλευτές, Λονδίνο, 21-24 Σεπτεμβρίου 2027 βουλευτές, ε, ετήσια συνέλευση του ΔΕΛΤΑΝΤΑΦ ε, Ουάσιγκτον 15-18 Οκτωβρίου, 7 βουλευτές και τέλος Λισαβόνα 4 και 5 Νοεμβρίου, 6 βουλευτές. Η κατανομή των εδρών θα συζητηθεί σε μια μελλοντική συνεδρίαση όταν υπάρξει η σχετική έγκριση των αποστολών δέκατων αναφορές, εγκρίθηκαν οι νέες κατευθυντήριες γραμμές, δίκτυο των αναφορών ζητήθηκε από του συντονιστέ να υποβάλουν τακτικά και αναπληρωματικά μέλη. Ακρόαση ΦΑΤΚΑ συμφωνήσαμε ότι η ΕΚΟΜ θα πρέπει να εμπλακεί στην οργάνωση μια δημόσια ακρόαση από την Επιτροπή Αναφορών. Ενδέκατο, δίκτυο ενσωμάτωση του φύλου. Ζητήθηκε από του συντονιστέ να υποδείξουν ονόματα για τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του δικτύου αυτού μέχρι τις 25 Οκτωβρίου. Επόμενο, τεχνικές συνεδριάσεις στο πλαίσιο τριμερών διαπραγματεύσεων. Εγκρίθηκαν οι κατευθυντήρες γραμμές ΕΚΟΝ μετά το αίτημα του συντονιστή του ECR. Συμφωνήθηκε ένας βοηθός ή ένας σύμβουλος αναμάδα να πηγαίνει στις τεχνικές συνεδριάσεις στο πλαίσιο των Εράνων ως παρατηρητής, χωρίς δικαίωμα λόγου. 13ο και τελευταίο ανακοίνωση για το ψήφισμα για το ΜΠΕΠΣ. Οι συντονιστές ενέκριναν το αίτημα της συντονίστριας των σοσιαλδημοκρατών για να υπάρξει ένα σχετικό ψήφισμα για το ΜΠΕΠΣ και την ψηφιακή φορολογία. Επίσης επιβεβαιώσαμε την οργάνωση μια ανοιχτή συνεδρίασή μας ε, μαζί με την ε, Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή της, ε, με την Κίνα και συμφωνήθηκε ότι η γραμματεία θα πρέπει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου να συντάξει ένα πίνακα με τις απαντήσεις που έχει λάβει η Κομισιόν στα διάφορα ζητήματα και εκθέσει πρωτοβουλία πρωτοβουλίας, μεταξύ των οποίων και το ψήφισμα ΚΟΜΕΞ. Και μετά οι συντονιστέ θα αξιολογήσουν. Αυτές ήταν λοιπόν οι ανακοινώσει. Το επόμενο θέμα είναι η έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων 24 Ιουλίου, 4 και 5 Σεπτεμβρίου, 16 Σεπτεμβρίου, 23-24 Σεπτεμβρίου, 2 Οκτωβρίου και 7 Οκτωβρίου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσει εγκρίνονται και Τώρα, επιτέλους, καλωσορίζω τους προέδρους των τριών θεσμικών οργάνων. Θα μας πείτε λοιπόν τι έχετε κάνει το τελευταίο έτος, ειδικά τον ρόλο σας στην συνεργασία με τους κανόνες, τον συντονισμό και την σύνταξη κανόνων. Να ακούσουμε επίσης ποιες είναι οι προτεραιότητες σας στους επόμενους 12 μήνες. Ο κύριος Μπερναρντίνο επίσης ε, θα μιλήσει και ως πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής ε, των ε, Τριών Εποπτικών Αρχών και θα μας πει πώς σκοπεύει να ασκήσει τα καθηκοντά του ως δεύτερος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Συστημικής Σταθερότητας. Ενημερώνω τους βουλευτές ότι οι τρεις πρόεδροι έχουν κάνει ήδη δηλώσεις οι οποίες έχουν δοθεί στους βουλευτές κάθε ε, πρόεδρος ε, του καθεσμικού οργάνου θα έχει δυνατότητα να κάνει κάποιες ε, παρατηρήσεις. Ο κύριος Μπερναρντίνο θα έχει συνολικά 10 λεπτά ως ε, πρόεδρος της Μεκτής Επιτροπής των Εποπτικών Αρχών και δεύτερος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ρυθμιστικής Σταθερότητας. Ο κύριος Καμπά και ο κύριος Μαγιόρ θα έχουν από 5 λεπτά. Μετά θα έχουμε ανταλλαγή απόψε με τους βουλευτές. Οπότε κύριε Μπερναρντίνο, έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκλησή σα και πάντα χαίρομαι να έρχομαι εδώ. Πρώτα απ' όλα ω πρόεδρο τη Μικτή Επιτροπή για, το... για τα τρία εποπτικά όργανα. Πρώτα απ' όλα θέλω όλους να σας συγχαρώ για τον ορισμό σας ή για τον επανορισμό σας στην Επιτροπή αυτή και την Πρόεδρο για την Προεδρία. Λοιπόν, οι τρεις ε, εποπτικές αρχές πάντα έχεραν τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και κυρίως των μελών της ε, ΕΚΟΝ και εννοείται ότι θέλουμε να έχουμε καλή συνεργασία μεταξύ μας. Τώρα, πού έχουμε καταλήξει και πώς έχει προχωρήσει το έργο μας στις τρεις αυτές υπηρεσίες. Να ξεκινήσω πρώτα από το σημαντικό μας έργο όσον αφορά την ε, διασταυρωμένη εποπτεία. Υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες βέβαια όσον αφορά την ε, απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν διάφορα σενάρια, υπάρχει το πιο ακραίο. Ε, Παρ' όλα αυτά, συνεργασία με τις Βρετανικές Αρχές ε, θα συνεχιστεί, τουλάχιστον αυτό είναι το μέλημα τη Μικτής επιτροπή. Θέλουμε επίσης να προλάβουμε ακραίες καταστάσεις και η Μικτή Επιτροπή περιλαμβάνει συστάσεις πολιτικής για θέματα μεταφοράς ε, βέβαια των οργανισμών. Επιπλέον, υπό το φως του σημερινού οικονομικού περιβάλλοντος και του σεναρίου που προβλέπει ακόμα χαμηλά επιτόκια, η Μικτή Επιτροπή εξετάζει διάφορες περιπτώσεις για τις οικονομικές υπηρεσίες προς όφελος των καταναλωτών. Εξετάζουμε επίσης και το ρόλο που μπορεί να παίξει το οικονομικό σύστημα για μια μεταβατική ε, μετάβαση αντιμετωπίζοντας όλες τις προκλήσεις. Τώρα, προστασία των καταναλωτών και καινοτομία. Βρίσκονται πάνω-πάνω στην ατζέντα της Μικτής Επιτροπής. Από τότε που ξεκινήσαμε με το έγγραφο KIT, που είναι το βασικό έγγραφο ε, πληροφοριών και τα PRIPS, οι υποπτικές αρχές έχουν δεσμευτεί να στηρίξουν την αποτελεσματική σύγκληση των κανόνων αυτών. Και γι' αυτό από το 2019 στείλαμε διάφορες ερωτήσεις και πήραμε απαντήσεις και κάναμε και διάφορες υποπτικές δηλώσεις. Είναι πολύ σημαντικά θέματα αυτά, τα οποία συζητήθηκαν όπως θα θυμόσαστε και είχαν θέσει πολλές ερωτήσεις εδώ στις 20 Φεβρουαρίου που μας πέρασε. Ε, τότε ακούσαμε τις ανησυχίες των διάφορων πλευρών όσον αφορά τους σημερινού κανόνες και είπαμε ότι θα φροντίσουμε να υπάρξει αναθεώρηση του κατεξουδότηση κανονισμού. Και χαίρομαι που μπορώ να σας ενημερώσω για τις εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα, έχουμε ε, αλλαγές όσον αφορά τα διάφορα ε, σενάρια επιδόσεων, το κόστος και τα πολλαπλά προϊόντα. Επίσης βασιζόμαστε και στο feedback βέβαια που έχουμε μετά από τις διαβουλεύσεις που έχουμε κάνει και από τις δοκιμές που κάναμε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πιστεύουμε ότι οι προτάσεις μας προσφέρουν να προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα όσον αφορά τον κανονισμό και την αναθεώρησή του και να προσφέρουμε στον καταναλωτή καλύτερα εργαλεία για να καταλαβαίνει καλύτερα και το kit θα μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα και διάφορα επενδυτικά προϊόντα όπως επίσης και τα use στα ΟΣΑΚΑ. Αυτό μπορεί να ενισχύσει βέβαια τη δυνατότητα των καταναλωτών να μπορούν να συγκρίνουν μεταξύ επενδυτικών προϊόντων και να υπάρχει ισότιμο πεδίο δράση για όλου. Επιπλέον, τον Ιούλιο 2019, η Μικτή Επιτροπή δημοσίευσε μια, ε, μια κοινή έκθεση ε, για διασταυρούμενη εποπτεία και αυτό βάσει διάφορων κανόνων passporting και λαμβάνοντας υπόψη τον εντοπισμό ε, των ε, αρχών που βασίζονται στην συνεργασία. Τώρα, ακολουθούμε και το πρόγραμμα της Επιτροπής, το πρόγραμμα δράσης για τα βιώσιμα οικονομικά. Και ε, τονίζουν αυτά ότι οι οικονομικές αγορές και όσοι συμμετέχουν, όπως επίσης και οι οικονομικοί σύμβουλοι, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους τους κανόνες που έχουν να κάνουν ναι, με το περιβάλλον, το κοινωνικό τομέα και τη διακυβέρνηση. Ο κανονισμός θα φροντίσει για την προστασία των επενδυτών ακόμα περισσότερο. Μπορούμε να έχουμε επίσης έξι τεχνικές προδιαγραφές σε επίπεδο προϊόντων. Επιπλέον θέλουμε να εντοπίσουμε την κατάλληλη μέθοδο για να αξιολογούμε και τις αρνητικές επιπτώσεις των ε, επενδυτικών αποφάσεων ε, επί των διώσιμων ε, παραγόντων. Το έργο μας αυτό συνεχίζεται. Τώρα, επίσης υπό τη Μικρή Επιτροπή έχουμε ετοιμάσει ένα νέο φόρουμ για τους διευκολυντές καινοτομίας και έχουμε έκθεση όσον αφορά το θέμα αυτό. Η έκθεση αυτή εντοπίζει την ανάγκη για δράση προκειμένου να υπάρχει καλύτερο συντονισμό και συνεργασία μεταξύ των διευκολυντών καινοτομία για να ε, βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την FinTech. Ε, υπάρχει πλατφόρμα λοιπόν για τους επόπτες να μπορούν να συναντιόνται τακτικά, να ανταλλάσσουν ε, απόψεις, να μιλούν με τις επιχειρήσεις, με τους διευκολυντές καινοτομιών και να καταλήγουν σε κοινή άποψη όσον αφορά τις υπηρεσίες, τα μοντέλα και την καταπολέμηση των απατών. Επιπλέον, τον Απρίλιο του 2019 οι ΕΣΕΣ δημοσίευσαν δύο γνωμοδοτήσεις ε, απαντώντας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο πρόγραμμα δράσης της για το FinTech. Μία έχει να κάνει με τις ε, τεχνολογίες ε, πληροφοριών και τους σχετικούς κινδύνους και η άλλη έχει να κάνει με τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο. Στόχος ε, των τριών υποπτικών αρχών είναι ότι κάθε σώμα πρέπει να υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες ώστε να προσφέρονται οι ρυθμιστικές υπηρεσίες ασφαλώς. Επίση, δουλέψαμε και όσον αφορά την νομοποίηση εισόδων παράνομες δραστηριότητες. Ε, Κυρίω επικεντρωθήκαμε σε στόχους που έχουν να κάνουν με σοβαρέ παραβάσεις και η Μικτή Επιτροπή επίσης ε, προχώρησε το έργο της για ε, ίδια πρωτοβουλία όσον αφορά τη συνεργασία για να υπάρξει ακόμα περισσότερη συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων διασυνοριακά. Επιπλέον, η Μικτή Επιτροπή το Σεπτέμβριο του 2019 εξέδωσε τη δεύτερη γνωμοδότησή της για την, τους κινδύνους από την νομοποίηση παράνομων εισόδων και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας μετά από τα μέτρα και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις προτάσεις της προκειμένου να υπάρχει σύγκληση και σε αυτό το τομέα. Τώρα ακριβώ επειδή η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών έχει αναλάβει και αυτό το έργο της καταπολέμησης, δηλαδή νομοποίησης προσόδων από παράνομες δραστηριότητες, θα προχωρήσει σε αυτό το έργο σε συνεργασία με τις άλλες δύο υποπτικές αρχές, τις οποίες θα συμβουλεύεται για τη συνέχεια του έργου. Τέλος, η Μεκτή Επιτροπή συνεχίζει το έργο της για τους χρηματοπιστωτικούς ομίλους και έχει διαβουλεύσει κάθε τόσο όσον αφορά τις διάφορες συναλλαγές και την ε, υπερβολική συγκέντρωση των ομίλων. Ε, φροντίζουμε να υπάρχουν προδιαγραφές και πλαίσια επίσης για τις ε, τη διάθεση στοιχείων από τους ομίλους αυτούς για να μην υπάρχει υπερβολική συγκέντρωση και ελπίζουμε να υπάρξει έτσι ισότιμο πεδίο δράσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έργο αυτό θα ολοκληρωθεί στα τέλη της χρονιάς αυτής. Συνεπώς κυρίες και κύριοι, θέλω να ολοκληρώσω τονίζοντας ότι η Μεκτή Επιτροπή θα συνεχίσει να επικεντρώνεται σε όλα αυτά τα σημαντικά θέματα και τα επόμενα χρόνια και προβλέπουμε σε επικοδομητικό και καρποφόρο διάλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ΣΕΣΕΚΟΝ. Τώρα επιτρέψτε μου παρακαλώ να περάσω στο θέμα της ΙΟΠΑ και στο έργο μας όσον αφορά την εποπτική σύγκληση και τις επιπτώσεις του οικονομικού σημερινού περιβάλλοντος στους διάφορους κλάδους. Θα επικεντρωθώ επίσης και στο κλίμα αυτή τον κίνδυνο στον κυβερνοχώρο κλπ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η εποπτική σύγκληση βρίσκεται στην καρδιά της δράσης μας. Στόχος μας είναι να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά την εποπτεία. Ε, τα τελευταία χρόνια είχαμε 11 διαφορετικές ε, πλατφόρμες, οι οποίες... Ε, Τύχε ένα συντονισμό από την ίδια την ΙΟΠΑ με επιχειρήσει οι οποίε πολλέ φορέ έχουν μοντέλα δράση τα οποία δεν είναι αρκετά ασφαλή. Όλα αυτά ε, τα διαπιστώσαμε κυρίως στον οικονομικό τομέα στην ε, Γαλλία και στην Ιταλία. Υπάρχουν διάφορες αποτυχίες, επτοχεύσεις επίσης και σε διασυνορικό επίπεδο που αποδεικνύουν ότι πρέπει να προστατεύσουμε πάρα πολύ την πολιτική μας και να υπάρξει ένα ε, δίκτυο με εγγυήσει, εναρμονισμένο όμως σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με επαρκή χρηματοδότηση. Επίσης, ενισχύουμε το έργο μας και για την εποπτεία των επιχειρήσεων. Έχουμε τέσσερις προτεραιότητες. Ε, ζωή, ζωής, πρώτα απ' όλα ε, πολλαπλά προϊόντα και ε, οι αξιώσεις όσον αφορά τα ατυχήματα, δυστυχήματα αυτοκινήτων. Εμείς έχουμε εντοπίσει διάφορα επιχειρηματικά μοντέλα τα οποία δεν είναι ασφαλή και απαιτούν περισσότερη εποπτεία. Και θα σας δώσω ένα μόνο παράδειγμα όπου τα νούμερα μιλάνε από μόνα τους. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν για κάθε 100 ευρώ που δίνει ο καταναλωτής για ε, ασφάλιση 77 πηγαίνουν κατευθείαν στο διανομέα και μόνο 14 επιστρέφουν κάποτε ως αξίωση στον καταναλωτή. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε εκδώσει και ε, οδηγίες όσον αφορά κυρίως τις ασφάλειες στον τομέα των ταξιδιών. Κάτι το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ τους καταναλωτές και μερικέ φορέ χρειάστηκε κάποια προϊόντα να αποσυρθούν από την αγορά. Όμω συνεχίζεται αυτό το αρνητικό περιβάλλον το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ και του καταναλωτέ, αλλά και του επιχειρηματίε. Θα έχουμε την αναθεώρηση το 2020 τη οδηγία Φερεγγιότητα 2 για να είναι πιο αποτελεσματική και να λειτουργεί καλά. Δεν αφιζητούμε βέβαια την βάση και τις εξελίξεις τις βλέπουμε σαν ε, πραγματικά κάτι θετικό και όχι σαν κάτι ανατρεπτικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην αναθεώρηση του 2018 της Solvency 2 δεν δέχτηκε τις προτάσεις μας. Οπότε ένα σημαντικό ζήτημα εδώ είναι η αναλογικότητα και η ΟΠΑ έχει κάνει προτάσεις για τη σημαντική μείωση των απαιτήσεων για ε, παροχή δεδομένων. Τα αποτελέσματα των δοκιμών που έγιναν το 2019 περιμένουμε ως αποτελέσματα όπου να είναι για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Τώρα, η κλιματική αλλαγή είναι επίσης κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε μια εκνομοδότηση φέτος για το πώς θα λάβουμε υπόψη μας τη Solvency 2 και τον κλιματικό παράγοντα. Θέλουμε στις κεφαλικές απαιτήσει να λάβουμε υπόψη μας την πράσινη διάσταση και θέλουμε και οι ασφαλιστές να συνεισφέρουν στην προσαρμογή και στη μετρίαση της κλιματικής αλλαγής μέσω επενδύσεων αλλά και μέσω των γενικότερων δραστηριοτήτων τους ε, ασφαλιστικών πρακτικών. Οι φυσικές καταστροφές τελευταία είναι πιο συχνές και πιο μεγάλες. Οι επιπτώσεις ε, ε, αυτών στις επιχειρήσεις και στο οικονομικό σύστημα είναι κάτι που δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε. Πιστεύουμε ότι η Ευρώπη πρέπει να δράσει μαζί για να ανταποκριθεί στην πρόκληση αυτή. Τώρα, όσον αφορά την ψηφιοποίηση και του κινδύνου στον κυβερνοχώρο, έχουμε αναθεώρηση όσον αφορά την άλυση των μεγάλων δεδομένων στην, ε, στα αυτοκίνητα και στην υγεία. Και εκεί φάνηκε ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ηθική στα ψηφιακά. Γι' αυτό και δημιουργήθηκε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων που θα βοηθήσει για την εφαρμογή των αρχών της ηθικής στο ψηφιακό κλάδο. Έχουμε όλο και περισσότερο εξελίξεις στην ε, ψηφιακή τεχνολογία, κάτι το οποίο θέτει νέες προκλήσεις. Θέλουμε να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις και θα γίνει αυτό με την ψηφιοποίηση, αλλά πρέπει να υπάρχει μια ε, στέρεα και υγιής τέτοια αγορά ώστε να μπορέσουν σε ανώνυμη βάση βέβαια να κυκλοφορούν τα δεδομένα αλλά με ασφάλεια. Τέλος, όσον αφορά την κεφαλαϊκή αγορά, εμείς πιστεύουμε ότι οι αποταμιευτές, οι ιδιώτες να μπορούν να υποφεληθούν από αυτή την αγορά και από τα κεφάλαια. Γι' αυτό και θέλουμε γρήγορη εφαρμογή των ΠΕΠ και πιστεύουμε επίσης ότι οι χώρες μέλη πρέπει να ενθαρρύνουν την συμμετοχή των συνταξιοδοτούμενων στα σχήματα αυτά και να βοηθήσουμε να υπάρξουν λύσεις οι οποίες είναι υγιείς και ασφαλές. Εν κατακλείδη, κυρίε και κύριοι, η ΟΠΑ θα συνεχίσει την αποστολή τη και θα αναλαμβάνει νέα καθήκοντα μετά από την ε, τελευταία αναθεώρηση με, με το βλέμμα κυρίω στα ζητήματα τα οποία έχετε θέσει εσεί. Θέλουμε να ικανοποιήσουμε τι προσδοκίε σα, γι' αυτό βέβαια χρειαζόμαστε πόρου, ανθρώπινου και οικονομικού και πιστεύουμε ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να στηριζόμαστε σε εσά. Εργαζόμαστε για μια Ευρώπη η οποία προστατεύει και η οποία δίνει νέες δυνατότητες. Θέλουμε μια οικονομία η οποία να λειτουργεί για τον άνθρωπο. Αυτό είναι και το μότο της Νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εννοείται είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσει. Ευχαριστούμε κύριε Μπερναρντίνο και τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Κάμπα. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ τη Οικονομική και Νομισματική Επιτροπή, κυρίε και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Είναι μεγάλη τιμή να εκπροσωπώ την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών στην πρώτη μου ακρόαση στην ΕΚΟΝ. Ε, πέρσι υπήρχαν πάρα πολλέ αλλαγέ στην Αρχή Τραπεζών και κυρίω ήταν η μετακόμιση μα Λονδίνο σε Παρίσι και δεύτερον. Ε, ε, είχαμε την εκλογή του Πρόεδρου και τελικά αρχίσαμε αυτή τη διαδικασία τον βρούμε ένα εκτελεστικό ε, διευθυντή Οπότε προχωρήσαμε σε όλα αυτά τα μέτωπα. Να σας πούμε αυτή την ευκαιρία τώρα τι έγινε. Ε, Ποια ζητήματα ήταν πάρα πολύ ε, σημαντικά για τους ε, εμπλεκομένους και ακριβώ για τον κόσμο. Όλα αυτά θα καθορίζουν την αποστολή μας. Ο τραπεζικός τομέας θωρακίστηκε περισσότερο. Αυτό είναι προϋπόθεση για να υπάρχει μια στιβαρή οικονομική ανάπτυξη. Οι ισολογισμοί επίσης έχουν γίνει πιο σταθερή στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά ε, και ε, τα κόκκινα δάνεια ε, πάνε τώρα καλύτερα, έχουν μειωθεί μισά από το 15, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να καταθέτουμε τα όπλα, θα πρέπει να προσέξουμε περισσότερο στο τι θα γίνει. Επίσης παραμένει μια πρόκληση το πώς θα υπάρξει περισσότερο κέρδος για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης να έχουμε μικρότερα περιθώρια όσον αφορά τις παραδοσιακές δραστηριότητες, αυξήθηκε το κόστος και μπορεί να αυξηθούν τα προβλήματα όσον αφορά την επιβράδυνση της οικονομίας σε διάφορες χώρες και όλα αυτά θα πρέπει να είναι προτεραιότητα για τις τράπεζες και ταυτόχρονα αυτές θα πρέπει να συνεχίσουν να ε, επενδύουν όσον αφορά τη διαχείριση κινδύνων και την τεχνολογικό μετασχηματισμό και έτσι να έχουμε πιο βιώσιμο πρότυπο οικονομίας τώρα ε, το stress test για το 2020 θα αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση το ολοκληρώνουμε και έτσι θα δούμε κατά πόσο μπορούν να αντέξουν τις ε, διαταράξεις ευρωπαϊκές τράπεζες και επίσης να δούμε πώς να βελτιώσουμε τα πράγματα στα stress test μακροπρόθεσμα και έτσι να μπορούμε να μειώσουμε το βάρος και την γραφειοκρατία για τράπεζες και εποπτικές αρχές και το να σας πω ποιες είναι οι προτεραιότητές μας. Θέλουμε να δούμε το τι θα γίνει με ε, την υλοποίηση της Τρίτης Συμφωνίας της Βασιλείας και να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ε, έχουμε ε, αντιμετώπιση των κινδύνων και θέλουμε γι' αυτό να υπάρξει μια μεταφορά των παγκοσμίων προτύπων σε κανονισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έτσι να είναι αξιόπιστο το νομοθετικό κανονιστικό μας πλαίσιο. Η αξιολόγησή μας ε, μας οδηγεί στο να δούμε τις επιπτώσεις στις ελάχιστες κεφαλουχικές απαιτήσει και επίση θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να απορροφηθεί από τις τράπεζες ε, στην μακρά περίοδο προσαρμογής. Οι επιπτώσεις για μικρομεσαίες τράπεζες είναι μικρότεροι, πιο συγκρατημένοι. Επίσης να δούμε μακροοικονομικά ποιες είναι οι επιπτώσεις. Θέλουμε να δούμε πώς θα υλοποιήσουμε όλες τις εντολές από το πρόσφατο πακέτο μέτρων για μείωση των κινδύνων και τα άλλα νομοθετικά ε, ζητήματα. Θέλουμε να υπάρχει χαρτής πορεία σε πολλούς τομείς, σε αμοιβέ, σε διακυβέρνηση, έκθεση εκτεταμένη, ε, δεύτερο πυλώνα και παράλληλα θέλουμε να συνεργαστούμε με την Κεντρική Τράπεζα και άλλα θεσμικά όργανα για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένο σύστημα για δεδομένα από πλευράς στατιστικής κλπ. Οπότε υπάρχει ένα σύστημα και να μας οδηγεί σε υποβολή εκθέσεων, σε αποκάλυψη υποχρεώσεων, σε συμμόρφες που να είναι πιο αποτελεσματικό και πιο εύκολο, οπότε τα χρηματοοικονομικά να είναι ε, βιώσιμα. Αυτό είναι στην καρδιά των στόχων μας και να δούμε πώς θα διευκολύνουμε τις τράπεζες για στρατηγική διακυβέρνηση και διαχείριση κινδύνων, οπότε θα πρέπει η έκθεση ε, σε όλα αυτά θα πρέπει να μελετηθεί αργότερα. Τώρα, ε, χρηματοοικονομική τεχνολογία ε, και καινοτομία θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μας δίνει την ευκαιρία για να έχουμε νέες τεχνολογίες που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα σε σχέση με νέες μορφές ανταγωνισμού και θα οδηγήσει σε ε, χρηματοοικονομική σταθερότητα. Μέχρι σήμερα έχουμε εκδώσει καθημερινές γραμμές για τις τράπεζες. Καλύτερη διακυβέρνηση, λιγότερη κίνδυνη όσον αφορά το outsourcing για το ε, νέφος, και επίσης τους ε, κινδύνους ICT με τα crypto assets και οπότε όλα αυτά θα βασιστούν στις ε, εμπειρίες μας από όλη την Ένωση για τις νέες τεχνολογίες, γι' αυτό έχουμε και αυτόν τον κόμβο σε σχέση με το FinTech στην Ευρωπαϊκή και ε, αυτό αφορά και την EFIF και επίσης άλλη αλλαγή προέρχεται γιατί έχει αλλάξει ο κανονισμός ο ιδρυτικός. Οπότε αυτό τώρα το ε, υλοποιούμε. Θα πρέπει να γίνει σεβαστή η διαφορετικότητα των ε, επιμέρους τραπεζικών δομών, αν υπάρχει αναλογικότητα, θα συγκροτήσουμε μια συμβουλευτική επιτροπή επί τη βάση του άρθρου 1.6 να καταπολεμήσουμε την διάθεση προϊόντος εγκλήματος. Αυτό είναι πρόκληση για όλη την Ευρώπη και αυτό φάνηκε από κάποιες διαβόητες ε, πρόσφατες υποθέσεις ο δε ιδρυτικός μας κανονισμός μας παρέχει ε, νέες αρμοδιότητες, το ώστε να παρακολουθούμε ε, και να χαράσουμε πολιτικές, να συντονιζόμαστε, να εποπτεύουμε. Έχουμε επίσης νέες αρμοδιότητες για μια καινούργια βάση δεδομένων, για εκτίμηση κινδύνων σε σχέση με τις ε, ε, εθνικές αρμόδιες αρχές όσον αφορά τους ε, επιμέρους παράγοντες του κλάδου. Οπότε θα έχουμε και μια διαρκή επιτροπή AML που θα εκπροσωπεί τις ε, αρχές από όλα τα κρατημέλη για να έχουμε συντονισμό και επίσης ε, θωρακισμένη, στεγανή εποπτεία για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και σας ευχαριστώ για αυτή την ευκαιρία που μας δώσατε και οπωσδήποτε και σήμερα αλλά και όποτε θέλετε θα σας παρέσχουμε διευκρινιστική Κύριε Κάμπο, ευχαριστούμε Πρόεδρος και τώρα το λόγο ο κύριος Μάγιορ. Συγγνώμη, συγγνώμη αν ε, πάμε λάθο το όνομά σα. Οπωσδήποτε το λέτε εσεί καλύτερα από ότι μιλάω εγώ Ιταλικά και είναι πολύ σωστό. Σας ε, ευχαριστώ λοιπόν. Κυρίες ε, και κύριοι βουλευτές, είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δίνετε να σας παρουσιάσω σύντομα τι δραστηριότητε της ΕΣΜΑ το τελευταίο έτος εν ώψη της νέας ε, θητείας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Γνωρίζω ότι για αρκετούς από εσάς ίσως αυτή είναι η πρώτη επαφή με την ΕΣΜΑ. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω με μια σύντομη εισαγωγή για την ε, αρχή μας και τον ρόλο που παίζουμε στις κεφαλαίες Η ΕΣΜΑ ιδρύθηκε το 2011 ως μια ανεξάρτητη αρχή και ο ρόλος της είναι να διασφαλίζει την προστασία των επενδυτών, την σταθερότητα και την εφταξία των αγορών. Αυτό γίνεται μέσω των τεσσάρων δραστηριοτήτων που έχουμε ανάπτυξη των ενιαίων κανόνων, η σύγκληση στον τομέα της εποπτείας, αξιολόγηση κινδύνων, αλλά και άμεση εποπτεία όσον αφορά τους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους και τα μέτρα σύγκλησης. Τα πρώτα χρόνια της ύπαρξή μας ε, αφιερώθηκαν στο να εφαρμόσουμε σωστά τις μεταρρυθμίσεις που ακολούθησαν την κρίση και τώρα αυξάνουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε την ίδια εποπτεία σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ανέφεραν και ο Γκάμπριελ και ο Χωσέ Μανουέλ. Για να στηρίξουμε λοιπόν το έργο αυτό που λέγεται Ένωση των Κεφαλαιαγορών θα πρέπει να ορίσουμε το σωστό ρυθμιστικό πλαίσιο και να διασφαλίσουμε το ότι οι κανόνες εφαρμόζονται σωστά και υπάρχει υποπτία στο εθνικό επίπεδο. Γι' αυτό ακριβώ θα ήθελα να σα πω το πώς σκοπεύουμε να εφαρμόσουμε τους στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζοντας την σταθερότητα και την προστασία των επενδυτών. Πρώτα απ' όλα, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, στον τομέα τη ε, βιώσιμη οικονομία, η ΕΣΜΑ έχει δώσει αρκετές τεχνικές συμβουλές στην Κομισιόν για το πώ διάφοροι συμμετέχοντε ε, στην αγορά, μεταξύ των οποίων και οι διαχειριστέ κονδολίων και οι επενδυτικές εταιρείες θα πρέπει να αξιολογούν τους παράγοντες της ε, αηφορίας για να αντιμετωπίζουν επαρκώς τον κίνδυνο του greenwashing. Κατόπιν οριστικοποιήσαμε τα στοιχεία των ε, κανόνων που αφορούν την τιτλοποίηση και τα σχετικά αποθετήρια τα οποία θα αποτελέσουν σύντομα αντικείμενο άμεσης εποπτείας μας. Και τέλος, επεκτείναμε τις λειτουργίες μας που αφορούν τα δεδομένα και την ανάλυση κινδύνου ενισχύοντας έτσι την διαφάνεια σε βασικούς ε, τομείς ε, προς όφελος των εποπτικών αρχών, ε, των πολιτικών και του γενικού, του ευρύτερου κοινού. Στο μέλλον λοιπόν θεωρούμε ότι έχουμε κάποια πράγματα ακόμα να κάνουμε και πρέπει να υπάρξει κάποια στοχευμένη δράση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους εθνικούς νομοθέτες και η ΕΣΜΑ θα τους στηρίξει όπου μπορεί είναι αυτή η τομής γενικά η χαμηλή συμμετοχή των νοικοκυριών και των μικροεπενδυτών στι δραστηριότητε των κεφαλαίων για να διασφαλίσουμε ότι τα νοικοκυριά θα έχουν καλύτερε αποδόσεις ε, στι αποταμιέσει του. θα πρέπει να επενδύσουν στις κεφαλαίε και όχι στι καταθέσει. Θα πρέπει λοιπόν να μειωθεί το σχετικά υψηλό κόστος των επενδυτικών προϊόντων όπως ανέφερε και η μελέτη μας. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερος ρόλος ε, των κεφαλαγορών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρώπης για να χρηματοδοτηθούν κοινοτόμες δραστηριότητες και να μειωθεί το επίπεδο χρέωσής τους. Ελπίζω να μπορέσουμε να συζητήσουμε σχετικές ε, πρωτοβουλίες τους μήνες που έρχονται. Το δεύτερο θέμα, το οποίο θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας, αφορά την εφαρμογή δύο πολύ σημαντικών ευρωπαϊκών νομοθετημάτων, τα οποία συμφωνήσαμε με την στήριξή σας, δηλαδή την αναθεώρηση των ε, εποπτικών αρχών και των emir 2.2. Θα ήθελα να παραλάβω την ευγνωμοσύνη μου προς την Επιτροπή σας που έχει παίξει σημαντικό ρόλο και μας εμπιστεύθηκε επιπλέον καθήκοντα και στην σύγκληση και στην εποπτεία και για να στηρίξουμε την ενιαία κεφαλαία αγορά, αλλά και για να έχουν οι κεφάλαια αγορές τα εργαλεία αυτά τα οποία είναι απαραίτητα καθώς αντιμετωπίζουμε και τον Brexit. Να σας ενημερώσω πως η εφαρμογή και των δύο κανονισμών βρίσκεται σε καλό δρόμο και αναμένουμε πως η υπηρεσία μας θα ξεκινήσει το 2020 να έχει πιο αποτελεσματικά εργαλεία για να επιτύχει την εποπτική σύγκληση, να εστιάσει περισσότερο στην προστασία των επενδυτών, να έχει νέε εσωτερικέ επιτροπέ μεταξύ των οποίων και μια επιτροπή αναλογικότητα και βελτιωμένη διοίκηση. Επίση, θα πρέπει να έχουμε τους πόρους ε, εγκαίρως για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε με τη νέα εντολή μας για τους κεντρικούς αντισυμβαλωμένους σύμφωνα με το ΕΜΙΡ 2 και αυτό αφορά και κάποιες τρίτες χώρες, τους λεγόμενους ε, αντισυμβαλωμένους της κατηγορίας 2. Ανέφερα ήδη επίσης ε, την σημασία που έχουν αυτά στην σύνθεση της νέας εποπτικής επιτροπής μας, όπως αναφέρει ο ΕΜΗΡ 2,2. Ήδη επίσης ανέφερα τον Brexit και θα ήθελα τώρα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις που αφορούν τον αντίκτυπό του στην δουλειά μας και στις ευρύτερες ευρωπαϊκές κεφαλαίες αγορές. Η ΕΣΜΑ έχει εργαστεί πάρα πολύ στην προετοιμασία του Brexit και χάρη στην εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με τις εθνικές αρμόδιες αρχές έχουμε επιτύχει ένα επίπεδο προετοιμασίας για ένα σενάριο Brexit χωρίς συμφωνία. Θα ήθελα να συμπενθυμίσω πως ε, λόγω του Brexit και τις διάφορες μετακομίσεις εταιριών συμμετεχόντων στην αγορά από το Ηνωμένο Βασίλειο, έχουμε ξεκινήσει ένα έργο ρυθμιστικής σύγκλησης με το δίκτυο συντονισμού, το οποίο μας έχει απασχολήσει σε πάνω από 230 περιπτώσεις εταιριών που μετέφεραν έδρα από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, ήθελα να καταλήξω υπογραμμίζοντας την σημασία της συνεργασίας μεταξύ της ΕΣΜΑ και της Επιτροπής σας. Από το 2011 το προσωπικό της ΕΣΜΑ αλλά και εγώ προσωπικά έχουμε αποδώσει μεγάλη σημασία στην επαφή με την Επιτροπή σας. Επίσης, εκτιμούμε τις πολλές ευκαιρίες που μας έχετε δώσει για να αναπτύξουμε τις απόψεις μας στα ζητήματα που εξετάζει η Επιτροπή σας. Ελπίζω πως ε, με την νέα σύνθεσή της η Επιτροπή σας και η ΕΣΜΑ να συνεχίσουν την συνεργασία αυτή με επικοδομητικό πνεύμα και στην Νέα Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Ερωτήσεις τώρα. Ισχύει πάντα ο κανόνα των πέντε λεπτών, δηλαδή δύο λεπτά ερώτηση και τρία λεπτά η απάντηση. Να είσαστε λοιπόν συνοπτικοί όσον αφορά τις ερωτήσεις. Αν είναι η ερώτησή σας προς έναν από τους τρεις προσκεκλημένους, παρακαλώ να το διευκρινίζετε. Εκ μέρους του ΕΛΚ, η κυρία Χούμπνερ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω συνεργαστεί με τον Στίβ Μέιερ τα τελευταία δύο χρόνια στενά, οπότε απλώς θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία αυτή και ελπίζω να ολοκληρώσετε το έργο σας στα ίχνη που ξεκινήσαμε δεν θα ρωτήσω εσάς κάτι, τον κύριο Μπερναντίνο θέλω να ρωτήσω, που δεν είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ μαζί του έτσι στενά. Οπότε θέλω να σας ρωτήσω για την ανταγωνιστικότητα του ασφαλιστικού κλάδου, γιατί ακούμε από εκπροσώπους του κλάδου ότι συνολικά ήμασταν αριθμός ένα, πάρα πολύ ανταγωνιστική, κάτι το οποίο δεν ισχύει πια, γιατί η Ασία έχει γίνει η πρώτη στη σειρά, έχει την πρώτη θέση. Ελπίζω να μην είναι αλήθεια, αλλά αυτά διαβάζουμε πάντως και αυτά ακούμε από τους εκπροσώπους του κλάδου. Τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια, ίσως ε, να το θυμόσαστε, ότι είχαμε συστήσει το θέμα της ικανότητας του ασφαλιστικού μας κλάδου να ανταγωνιστεί διεθνώς με τις εταιρείες που έρχονται από νομολογίες με εντελώς διαφορετικές ρυθμίσεις και καθεστώτα. Τώρα λοιπόν ε, δημοσιεύσατε αυτή την ε, καλή πρόταση για την αναθεώρηση της οδηγίας Φερικιότητα 2. Μπορείτε να σχολιάσετε παρακαλώ για τον αντίκτυπο που θα έχει η πρότασή σας στην ανταγωνιστικότητα του ασφαλιστικού κλάδου παγκοσμίω. Απάντηση του κ. Μπερναρντίνο. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Βεβαίως, ευχαρίστως να έχουμε πιο στενή συνεργασία μαζί. Τώρα να σας πω δύο λόγια για το θέμα της ανταγωνιστικότητας. Οι ασφαλίσεις είναι από τους κλάδους της οικονομίας όπου οι ευρωπαϊκές εταιρείε θα έλεγα ότι έχουν πολύ σημαντική θέση διεθνώς. Όπως βέβαια είπατε και είναι σωστό, έχουμε τώρα ασιατικές επιχειρήσεις που ανεβαίνουν πολύ, κυρίως βέβαια στην Ασία, όπου ο πληθυσμός αυξάνει με ταχύτατους ρυθμούς και τα νούμερα παίζουν ρόλο στον ασφαλιστικό κλάδο. Πάντως οι ευρωπαϊκές εταιρείες και χάρη στις αλλαγές που έγιναν με την οδηγία Φερεγγιότητα 2, με τις διάφορες πρακτικές, με πιο σύγχρονο καθεστώς, διατηρούν καλή τη θέση τους διεθνώς. Βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι διεθνώς θέλουμε να υπάρχουν ίδιες προδιαγραφές παντού όπως υπάρχουν ε, και στην Ευρώπη. Μένει πολλή δουλειά να γίνει. Έχει ήδη γίνει βέβαια τα τελευταία χρόνια ώστε να δημιουργηθούν ε, προδιαγραφές παγκοσμίως που να προσφέρουν ισότιμους όρους ε, δραστηριότητας. Όχι όσον αφορά τις κεφαλακές απαιτήσει ίσως, αν έχουμε πάντω τι ίδιες προδιαγραφέ στην Ευρώπη, στην Ασία και αλλού, αυτό θα βοηθούσε πολύ. Νομίζω ότι σε δύο εβδομάδε θα έχουμε περισσότερα νέα για τι εξελίξει όσον αφορά τι προδιαγραφέ αυτέ για τι κεφαλαικέ απαιτήσει. Τώρα για την αναθεώρηση τη Solvency 2. Θα σα πω που βρισκόμαστε. Ουσιαστικά ολοκληρώσαμε, θα έλεγα, το πρώτο στάδιο της διαδικασίας. είχαμε έναν μεγάλο κατάλογο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς αναλύσαμε προσεκτικά τις τεχνικές πτυχές. Ήδη από τον Ιούλιο έχουμε δημοσιεύσει κάποια συμβουλευτικά έγγραφα και συνεχίζουμε και τώρα. Υπάρχει διαφάνεια πάντως. Είμαστε πολύ ανοιχτοί για διάφορες επιλογές και τεχνικές επίσης επιλογές. Τώρα είμαστε στο δεύτερο στάδιο, αρχίζουμε τώρα της διαδικασίας, για να δούμε συνολικά το θέμα. Και όπως είπα και στην παρέμβασή μου, δύο θέματα είναι για μας σημαντικά. Το ένα είναι τα χαμηλά επιτόκια, που βέβαια πρέπει να αντικατοπτρίζονται με καλύτερο τρόπο στην αναθεώρηση της φερεγγιότητας 2. Γιατί ξέρουμε τι σημαίνει να έχει κανείς αρνητικές αποδόσεις. Οπότε αυτό σίγουρα θα πρέπει να το δούμε. Αλλά πέρα από αυτό, θέλουμε να κάνουμε πρόταση για ε, ισορροπή και ισότιμη κατάσταση όσον αφορά τον αντίκτυπο. Δεν είναι μόνο το ε, να υπάρχουν περισσότερα κεφάλαια. Δεν μπορεί από μια μεριά να έχουμε ε, πάρα πολλά κεφάλαια και από την άλλη να μην έχουμε αρκετά. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Και το τρίτο στάδιο θα είναι ακριβώς γι' αυτά του χρόνου, το πρώτο τρίμηνο, θα έχουμε μια συνολική αξιολόγηση αντικτύπου. Θα δούμε δηλαδή όλα τα μέτρα συντονισμένα για να δούμε ποιος θα είναι ο αντίκτυπος στον κλάδο. Και θέλουμε κάτι ισορροπημένο, όπως σας είπα, για να είναι ακριβώς σε καλή θέση και εύρωστος ο κλάδος. Ευχαριστούμε. Τώρα ο κύριος Φερνάντες, εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Καλησπέρα. Ισπανικά θα μιλήσω και ρωτάω τον πρόεδρο της ΕΣΜΑ, τον κύριο Μαϊόρ. Στην παρέμβασή σας είπατε ότι πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή αναλογικότητας στα πλαίσια της ΕΣΜΑ, αν κατάλαβα καλά αυτό που είπατε. Πολλές φορές τα επιχειρήματα υπέρ της αναλογικότητας ε, γενικά είναι αποδεκτά, αλλά μερικές φορές δημιουργούν κενά στη ρύθμιση. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πιο συγκεκριμένα. Τι αποστολή έχει αυτή η Επιτροπή Αναλογικότητας που προτείνεται να δημιουργηθεί τους επόμενους μήνες. Δεύτερη ερώτηση. Για άλλα κενά τρύπες στην εφαρμογή της σημερινής εποπτείας λέτε ότι πρέπει να βελτιωθεί η εποπτική σύγκληση με τις εθνικές εποπτικές αρχές. Και δεδομένου το θέμα είναι πολύ σημαντικό, κυρίως στα πλαίσια της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου του χρόνου, θέλω να ξέρω ποια είναι η κατάσταση, πόσο σοβαρή είναι η διαφοροποιημένη εφαρμογή της εποπτείας στις διάφορες χώρες μέλη γιατί στην έκθεση που δημοσιεύσατε και μας παρουσιάσατε αναφέρονται διαφορετικά σενάρια, MIFID, MIFID 2 και η εποπτεία αυτή δημιουργεί κάποια κενά γεωγραφικά. Πόσο σοβαρή είναι αυτή η κατάσταση ότι δηλαδή δεν υπάρχει εποπτική σύγκληση. Ευχαριστώ για την ερώτησή σας. Ας αρχίσουμε με το θέμα του κινδύνου και το Brexit. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μια ενσωματωμένη ε, κεφαλαϊκή αγορά, με βέβαια διαφορετικά σημεία εισόδου και με έναν ρυθμιστή έχετε πρόσβαση στην ευρωπαϊκή κεφαλαία αγορά. Τώρα η ερώτηση είναι σε τι βαθμό οι εθνικοί ρυθμιστές στο σημείο που βρίσκονται κάποια προϊόντα τα οποία πολλούνται διασυνοριακά. Τι συνέπειες μπορεί να έχουν τα προϊόντα αυτά σε άλλα σημεία της Ευρώπης. κατά πόσο δηλαδή αυτό λαμβάνεται υπόψη από τον ρυθμιστή στη συγκεκριμένη χώρα μέλος. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την ίδια τη δημιουργία των εποπτικών αρχών. Το 2011 στην έκθεση Λαροαζιέρ αναφερότανε αυτό το θέμα του ανταγωνισμού. Και με το Brexit, όπως καταλαβαίνετε, οι συμμετέχοντες από την αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου μετακομίζουν στην υπόλοιπη Ευρώπη, Οπότε το ερώτημα είναι, οι ρυθμιστές αυτοί εφαρμόσουν τις ίδιες προδιαγραφές παντού στην ε, Ευρώπη. Εννοείται ότι αυτοί που μας έρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο θέλουν να διατηρήσουν όσο γίνεται μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων του στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ενώ οι υπόλοιποι 27 θέλουν να έχουν 27 τη δυνατότητα και εποπτείας αυτών των ε, νεοφερμένων. Πώς το αντιμετωπίζουμε αυτό? Συμφωνία με τα διάφορα διεκτικά συμβούλια, ώστε ε, οι οργανισμοί αυτοί που έρχονται στην Ευρώπη να συζητούν με την ΕΣΠΑ ποια είναι τα ελάχιστα που πρέπει να τηρούν ώστε ο εθνικός ρυθμιστή να δούμε πώς μπορεί να τα λάβει αυτά υπόψη του. Και συμφωνήσαμε και για μια αξιολόγηση μεταξύ ομοτήμων για να δούμε κατά πώς, πώς έχουν λειτουργήσει τελικά αυτές οι μετακομίσεις. Τώρα για το θέμα της αναλογικότητας. Έρχεται στα πλαίσια της αναθεώρησης. Δεν πρόκειται μόνο για την ΕΣΠΑ εδώ, πρόκειται και για τις άλλες δύο εποπτικές αρχές. Ε, που συμμετέχουν στην ε, Επιτροπή αυτή αναλογικότητα. Συζητάμε μαζί τη μορφή της. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είναι μια επιτροπή η οποία ex θα βλέπει πόσο επιτυχώς ελήφθη υπόψη η αναλογικότητα. Γιατί τώρα όταν ε, κοιτάμε τις προδιαγραφές, κάνουμε την ανάλυση βέβαια κόστους ωφέλους και πολύ σωστά εσείς λέτε ότι η αναλογικότητα δεν πρέπει να είναι επιχείρημα για να πέφτουν οι προδιαγραφές. Όταν υπάρχει μια δραστηριότητα ε, που λαμβάνει η χώρα μέσω ενό πιο μικρού φορέα, ε, πρέπει να φροντίσουμε να είναι ισότιμη κατάσταση μεταξύ μικρών και μεγάλων. Ευχαριστώ. Ρινιού. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Έχω δύο ερωτήσεις για τον κύριο Κάμπα. Λέει Γαρικάνο. Ανησυχούμε σοβαρά όσον αφορά το θέμα της καταπολέμησης ε, της διάθεσης προϊόντων εγκλήματος και εσείς μας είπατε ότι η αρχή τραπεζών, η EBA, ε, έχει ε, κάποιο πρόβλημα σε ανθρώπινους και υλικούς πόρους. Βέβαια, με την ευκαιρία που ήρθατε εδώ, μας λέτε ότι υπάρχει δέσμευση για ένα νέο φορέα μια που τώρα λοιπόν το έχετε αυτό, κάποιες ε, χώρες μέλη θέλουν να υπάρχει μια τέτοια υπηρεσία, ανεξάρτητη αρχή ε, κατά Νέα υπηρεσία με αρμοδιότητες ουσιαστικές όσον αφορά την παρέμβαση ε, σε αυτό το μέτωπο, στα κράτη-μέλη. Εσείς τι θέση έχετε όσον αφορά το κατά πόσον χρειάζεται μια νέα υπηρεσία και πώς θα πρέπει αυτή να είναι διαρθρωμένη ούτως ώστε να συμπληρώσει το έργο της δικής σας υπηρεσίας Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Κάτι άλλο τώρα σε σχέση με την ε, εναλλαγή των αξιωματούχων σε διάφορες θέσεις. Τι γίνεται με το λόμπι των ε, χρηματοοικονομικών αγορών και εσάς. Καταλαβαίνετε ότι είναι εύλογη η ανησυχία μας τι μέτρα θα υπάρξουν ούτω ώστε να μην έχουμε συγκρούσεις συμφερόντων που είναι προφανές ότι θα προκύψουν. Δεν καταλαβαίνω κάποιες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Τραπεζών. Οπότε εμείς θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να συναντώμεθα με τον κύριο Φάρκας για αυτόν τον λόγο με χρυσό του αποφασίσουμε κάτι σε σχέση με αυτό το θέμα το οποίο αποτελεί σημαία του λαϊκισμού. Βεβαίως και υπάρχουν κάποιες κατα... καταστάσεις που δεν δημιουργούν συγκρούσεις συμφερόντων, αλλά προκειμένου υπάρχει το πρόβλημα. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό. Ο επόμενος. Ο κύριος Κάμπα. Πώς αφορά τον κανονισμό EML, για την Ευρωπαϊκή Ένωση αρχές Σεπτεμβρίου τα συζητήσαμε και ε, χαίρομαι που ήρθα να σας πω τις θέσεις μας. Αυτός ο κανονισμός βασίζεται στις σχετικές οδηγίες. Και βέβαια υπάρχουν πολλές απόψεις για το πώς ε, θα υλοποιηθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το θέμα είναι να υπάρχει αποτελεσματικός συντονισμός. Άρα ευτυχώς που το Κοινοβούλιο έδεσε αυτό το ζήτημα στην Νέα Επιτροπή, η οποία θα πρέπει να το συζητήσει. Τώρα για το τι θα κάνουμε. Έχουμε μια σειρά επιλογών. Πρώτο βήμα είναι το να υπάρξει κοινή προσέγγιση με τον κοινό κανονισμό. Να έχουμε μια προσέγγιση επί τη βάση της μεθόδου της οδηγίας. Άρα, ε, λιγότερο βάζουμε σε γενικές αρχές και περισσότερο σε κατευθυντήριες γραμμές. Αλλιώς δεν μπορεί να υπάρχει ε, μια ομοιογενής πολιτική παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν διαφορετικές πρακτικές. κοινή κανονισμή, κοινέ εποπτικές ε, πρακτικές και από την άλλη μεριά υπάρχουν διαφορετικές νομικές παραδόσεις όσον αφορά την προσφυγή στη δικαιοσύνη. Οπότε δυσκολεύονται τα πράγματα. Είναι θέμα συνεργασίας δικαστικών αρχών, διοκτικών αρχών, Γι' αυτό είναι δύσκολη η κοινή προσέγγιση. Όμως, κοινή υποπτία, κοινά πρότυπα, κοινή αξιολόγηση, αυτό οδηγεί σε περισσότερο ομοιογενή υλοποίηση. τρόσου να αφορά τον εκτελεστικό διευθυντή, είπαμε ότι ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από την EBA. Από την αρχή είπαμε ότι υπάρχει θέμα σύγκρουσης συμφερόντων με την ανάληψη των καθηκόντων του και η επιτοπτική επιτροπή που ασχολείται με αυτά για το διεδικό μας Συμβούλιο ασχολήθηκε και είπαμε ότι υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί από τη στιγμή που ανακοίνωσε την ανάληψη των καθηκόντων του εμείς είπαμε να υπάρξει η μεγαλύτερη διπροβλημόνη παρένθεση του ΣΥΠΗΝ των έξι μηνών. 2 Αυγούστου είπε ότι θα φύγει και άλλοι περιορισμοί δεν του επιτρέπεται να έρθει σε επαφή με οποιονδήποτε στην αρχή τραπεζών για οποιοδήποτε θέμα πολιτική μα δύο χρόνια αφού φύγει μέχρι δηλαδή το 2022 το Φεβρουάριο 18 μήνες δεν μπορεί να συνεργαστεί με οποιοδήποτε πεινάβουμε και για οποιοδήποτε από τα θέματα στα οποία έχει εργαστεί τα τελευταία τρία χρόνια. Χαίρομαι που θέσατε το ζήτημα. Οπότε, δεν έχει ανακατευθεί σε κανένα θέμα μας, σε καμία πολιτική μας και είπαμε και σε όλο το προσωπικό ότι δεν πρέπει να έχουν επαφή μαζί του και αν έχουν να απευθυνθούν στην Επιτροπή Ελέγχου Συγκρούσεων Συμφερόντων. Πρόκειται για 18 μήνο περιορισμό. Δεν μπορεί να ασχοληθεί με τίποτε επί 18 μήνες από σε όσα θέματα έχει ασχοληθεί ως υπάλληλος της EBA. και εσείς δικαιούστε να κάνετε αυτό το οποίο είπατε και είναι και το σωστό από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις εξηγήσει. Ε, τώρα ο κύριος Γιουνούς από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Για και Λούνες, με συγχωρείτε. Θα ήθελα να ρωτήσω τον πρόεδρο της ε, κοινή Επιτροπής. Με βάση την παρουσία σας εδώ πέρα, αναφέρατε την ανάγκη να υπάρξει μια ρυθμιστική σύγκληση στον τομέα της ασφάλειας αλλά και σε άλλους ε, τομείς ε, προφανώς ο συναδελφός ανέφερε τον ε, ρυθμιστικό ανταγωνισμό ως πρόβλημα και το βλέπω και στη χώρα μου αυτό. Στο έγγραφο εδώ πέρα από διάφορους που είχαν σχέση με την τράπεζα διεθνών διακανονισμών. Αναφέρονται διάφορα μοντέλα τα οποία θα αναφέρω. Έχουμε ένα μοντέλο κλαδικό, ολοκληρωμένο ή το λεγόμενο Twin Peaks των δύο κορυφών. Οπότε υπάρχει εδώ πέρα μια άνομη ομορφία παγκοσμίως και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με βάση και την δική σας εμπειρία και των συναδέλφων σας. Παραδείγματος χάρη είχε έρθει εδώ πέρα ο κύριος Ντομπρόφσκης ε, και είπε να έχουμε ένα μοντέλο με δύο κορυφές το οποίο ζήτησε επίσης και το γνωστό Ινστιτούτο Μπρέγκελ. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα, όπως ξέρετε, ε, σύγκρουση συμφερόντων. Ε, επίσης απαιτούνται διαφορετικές δεξιότητες για την εποπτεία της συμπεριφοράς και την ε, προληπτική υποπτία. Λοιπόν, δεν μπορούμε να έχουμε μια αποτελεσματική ενιαία αγορά χωρίς να υπάρχει μια ενιαία υποπτική υποδομή και σύστημα. Ποια είναι η απόψή σας? Έχετε κάποια προτίμηση προς κάποιο από αυτά τα μοντέλα ή ένα μοντέλο με τρεις κορυφές ίσως, γιατί βεβαίως υπάρχει και το θέμα του οικονομικού εγκλήματος. Οπότε ίσως θα πρέπει να σκεφτούμε με τρόπο πρωτότυπο πέρα από τα υφιστάμενα μοντέλα. Ποια είναι η άποψή σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πράγματι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση αυτή. Μπορώ να σας δώσω την ε, προσωπική μου άποψη όσον αφορά την ε, εμπειρία που έχω άλλωστε από ε, την εμπειρία μου, την εργασία μου ψηρά ετών. Θεωρώ πραγματικά ότι δεν υπάρχει κάποιο μοντέλο το οποίο μπορεί να καθοριστεί ως προτιμητέο από τα υπόλοιπα. Αν δούμε τις διάφορες ε, κρίσεις ε, που έχουμε, δεν υπήρχε κάποιο μοντέλο το οποίο αποδείχτηκε τελείως ε, θωρακισμένο. Διαφορετικές χώρες σε διαφορετικές περιπτώσεις είχαν αποτελέσματα με διαφορετικά μοντέλα. Οπότε, για να είμαι ειλικρινής, ε, δεν θεωρώ ότι υπάρχει ένα μοντέλο που μπορεί να θεωρηθεί ότι υπερέχει από τα υπόλοιπα. Αυτό το οποίο βλέπω ότι είναι σημαντικό είναι να φροντίσουμε ανεξαρτήτως μοντέλου που ακολουθείτε να υπάρχουν κάποια θεμελιώδη στοιχεία που θα αποτελούν κομμάτι της ε, εποπτείας στις διάφορες ε, χώρες και αναφερόμενο σε ένα ζήτημα που θίξατε κι εσείς. Η εμπειρία μου τα τελευταία χρόνια πηγαίνει προς την κατεύθυνση ότι βεβαίως υπάρχουν διαφορές στον τρόπο άσκησης της προληπτικής ε, εποπτείας, ειδικά στον τομέα της ασφάλειας και των συντάξεων και έχουμε πλέον μια πιο κοινή προσέγγιση, αλλά βεβαίως οι προκλήσεις είναι ακόμη μεγαλύτερες και εκεί πέρα θεωρώ ότι πρέπει να ρίξουμε μεγαλύτερο βάρος ως Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί Έχουμε και τα τελευταία χρόνια διάφορα νομοθετήματα που ακριβώς ρίχνουν μεγαλύτερο βάρος στην προστασία των καταναλωτών και τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και συχνά ήμουν πολύ ομόσος προς αυτό. Δηλαδή τα πάμε πολύ καλά με το να γράφουμε κανονισμούς ε, στην Ευρώπη, συλλογικά μέσω Συμβουλίου, Κοινοβουλίου, Κομισιών, Ευρωπαϊκών Αρχών, Εθνικών Αρχών, ε, ενδιαφερομένων. Νομίζω ότι παράγουμε καλούς κανονισμούς. Δεν είμαστε όμως εξίσου καλοί στην εφαρμογή και στην ε, επιβολή. υπάρχουν διάφοροι τομεί επίσης όπως παραδείγματο χάρη η εναλλακτική επίλυση διαφορών που αναφέρατε πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερο βάρο στην εφαρμογή μεγαλύτερη σύγκληση και συνοχή και στο να διασφαλίσουμε ότι θα πρέπει να είναι προτεραιότητα ακριβώ ε, το να λειτουργούν οι επιχειρήσει. γιατί αυτό έχει σημασία, να υπάρχουν αποτελέσματα για του ε, πολίτε. Ε, να έχουν προϊόντα τα τα προϊόντα τα οποία αγοράζουν να έχουν κάποια στοιχεία βεοντολογικά ε, και τα σχετικά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ευρωπαϊκή προσέγγιση αντί να έχουμε μία ενιαία αρχιτεκτονική σε ολόκληρη την Ευρώπη όσον αφορά την εποπτεία. Σας ευχαριστώ για το ID Αντώνιο Ρινάλντι. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λοιπόν, οι ερωτήσει ουσιαστικά αφορούν τον πρόεδρο, τον κύριο Κάμπα. Βλέπουμε εδώ πέρα μια διακριτική μεταχείριση εις βάρος των εμπορικών τραπεζών της Ένωσης που ουσιαστικά υποστηρίζουν την πραγματική οικονομία και το παραγωγικό σύστημα. Αντιθέτω, οι επιχειρήσεις οι οποίες δρούν κυρίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα είναι όμως ε, εκτεθειμένες σε πάρα πολλούς ε, μεγάλους ε, κινδύνους οι οποίοι δεν έχουν αρκετή εποπτεία και μπορούν να αποσταθεροποιήσουν ολόκληρο το τραπεζικό σύστημα. Επίσης διάφοροι φόβοι γίνονται από τους υψηλούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν διάφορα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι ζημιές που έχουν από τα διάφορα asset που έχουν και αφορούν ακριβώς αυτά τα οποία αναγράφονται στο κεφάλαιο 11.3 αφενός ε, και από τους κεντρικούς ε, αντισυμβαλόμενους και από τον κανονισμό ΕΜΙΡ. Υπάρχει βεβαίως ε, ιδιαίτερος ο κανονισμός 648 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, η EBA δεν θα έπρεπε να αναπτύξει κάποιες κατευθυντήριες γραμμές με συγκεκριμένες μεθοδολογίες για να μειώσει αυτούς τους κινδύνους που μπορούν να αποτελέσουν συστημικό κίνδυνο, καθώς μιλάμε για μεγάλες ευρωπαϊκές ε, τράπεζες. Και τέλος έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία να ελέγξουμε εάν ε, το κεφάλαιο αυτό των ε, τραπεζών αυτών σε σχέση με τις ε, υποχρεώσεις τους ε, επαρκεί για να ε, ανταποκριθεί σε περιπτώσεις κραδασμών. Λαμβάνοντας υπόψη πως τα λεγόμενα μη εξυπηρετούμενα δάνεια υφίστανται, σε, υφίστανται πολύ περιοριστική μεταχείριση και έτσι έχουμε έναν υπολογισμό αυτών των κινδύνων με μια αυτοαναφορική λειτουργία των τραπεζών. Τέλος, θα ήθελα να γνωρίζω πώς σκοπεύει να κινηθεί η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή όσον αφορά τις τεχνικές αρχές για την κατάρτιση software όπως προβλέπει το νέο άρθρο 36 του κανονισμού για τις κεφαλαιακές απαιτήσει που έχει ως ε, προθεσμία τον ε, Ιούνιο του 2020. Αλλά το ζήτημα είναι κατεπήγον γιατί οι ευρωπαϊκές ε, τράπεζες έχουν μειονέκτημα σε σχέση με τους Αμερικανούς ανταγωνιστές τους, αλλά και τις μη τραπεζικές επιχειρήσεις. Σας ευχαριστώ. Thank you. Thank you for the question. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. και θα αρχίσω με τους μεγάλους, πιο περίπλοκους οργανισμούς. Όπως ξέρετε, οι σχετικοί κανονισμοί είναι συστημικοί και συμπεριλαμβάνονται στην νομοθεσία που αφορά ε, τη συνολική συστημική προστασία που συμπληρώνουν την εθνική αντίστοιχη που υπάρχει ήδη έτσι κι οι οργανισμοί αυτοί υποβάλλονται σε κανονισμούς και στην ε, προστασία που ήδη προβλέπεται σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον, για τους κινδύνους της αγοράς από το 2012 και μετά έχουν γίνει πάρα πολλά προκειμένου να μην υπάρχει τέτοια έκθεση ε, των τραπεζών, είναι οι αντισυμβαλόμενοι, είναι η νέα νομοθεσία Βασιλεία 3 και άλλες ρυθμίσεις που έρχονται και θα έχουμε και στο τέλος αυτού του μήνα και που πιστεύουμε ότι πρέπει να εφαρμόζονται παντού. Είναι σημαντικά όλα αυτά και εκτιμήσεις μας για τις μεγάλες συστημικές τράπεζες και τις κεφαλικές απαιτήσει είναι της τάξης του 2%. Οπότε υπάρχουν αυτά τα μέτρα. Τώρα για τα MPLs, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, οι τράπεζες έχουν μειώσει κατά πολύ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τους τελευταίους μήνες, μερικές φορές και στο 50%. Η προσπάθεια βέβαια πρέπει να συνεχιστεί, κυρίως σε νότιες χώρες όπου συνεχίζουν να είναι μεγάλα τα ποσά και πολλά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Έχουμε και το πρόγραμμα δράσης για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έχουμε διαβούλευση αυτή την εποχή και κατευθυντήριες γραμμές για να δούμε πώς θα λαμβάνονται υπόψη. Για την τελευταία σας ερώτηση έχουμε ρυθμιστική εντολή για να εκτιμήσουμε την κατάσταση που επικρατεί Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ξέρουμε ε, ποιο, ποια είναι η τιμή, πόσο είναι το ποσό δηλαδή αυτών ε, αυτού του χρέους, του δημόσιου χρέους. Έχουμε πάντως διμερώς συνομιλίες με πολλές τράπεζες. Μας στέλνουν δεδομένα, εμείς επιστρέφουμε με νέες ερωτήσεις, ανακατηγορία και υπάρχουν και τεχνικές προδιαγραφές βέβαια που πρέπει να εφαρμόζονται και να συνοδεύουν την εθνική νομοθεσία. Να υπάρχουν δηλαδή κάποια προγράμματα για την εποπτική προστασία. Ελπίζω να έχουμε περισσότερα του χρόνου. Πρόεδρο, σε ευχαριστούμε. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Άτινγκ από το ECR, θέλω να σας υπενθυμίσω ότι έχουμε λιγότερο από 10 λεπτά στη διάθεσή μας. Α, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Λάθος. Έχουμε χρόνο, έχουμε χρόνο. Εγώ έκανα λάθος. Α, και είπα από όπου. Εντάξει, ευτυχώ, τρόμαξα. Ωραία, παρακαλώ κύριε Άτκιν. Όχι, μην τρομάστε. Επιτρέψτε μου να μιλήσω ολαδικά και να ρωτήσω κάτι στον κύριο Μαγιόρ. Οπότε θα μιλήσω τη γλώσσα μας. Κύριε Μαγιόρ, σήμερα διάβασα στο σταθμό του Ρότερνταμ παρακολούθησα και ένα interview δικό σας όπου λέτε ότι πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση όσον αφορά τις ε, ομολογίες. Και υπάρχουν προβλήματα που μπορεί να δημιουργήσουν κινδύνους για τη σταθερότητα του οικονομικού συστήματος. Ε, δεδομένου και του Brexit, και έτσι αλλιώς υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι εξαιτία του Brexit της τάξης των 10 ε, δισεκατομμυρίων. Αυτό που βρίσκω ότι είναι πολύ σημαντικό είναι να υπάρχει μια επεκτατική ε, πολιτική από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ώστε οι ε, επενδυτές οι οποίοι έχουν χαμηλές αποδόσεις να μην πέσουν και στον κίνδυνο αυτών επιπλέον. Οπότε εσείς μπορείτε να μας δώσετε κάποιες ενδείξεις για το τι κάνουμε με τον κίνδυνο αυτό του οικονομικού συστήματος, πώς τον απορροφούμε, τι συγκεκριμένα μέτρα παίρνει η ΕΣΜΑ ή θα πάρει και μάλιστα σε συνδυασμό με τους εθνικούς ε, επόπτες για να προστατεύονται ε, τα ποσά τα οποία επενδύονται και τις δύσκολες, δύσκολα διαχειρίσιμες επενδύσεις. Το πρόβλημα βέβαια είναι ο αντίκτυπος της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία μόνο φούσκες δημιουργεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, παντού, με δηλητηριώδη τελικά ε, προϊόντα το οποίο δημιουργούν περισσότερα προβλήματα παραλύσεις. Οπότε, κύριε Μαγιέρα, εσείς που είσαστε επόπτης, δεν έχετε καθήκον τις νομισμαστικές μας αρχές, τον πρόεδρο Τράγκη που έφυγε και τον αποχαιρετήσαμε με την Πανοκρισίες, δεν θα έπρεπε να μας προστατεύσετε από μια τέτοια νομισματική πολιτική. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πίνγκ. Και ευχαριστώ πολύ. Ωραία, Ολλανδικά. Α, μιλήσατε εσείς, αλλά νομίζω ότι και με τα αγγλικά θα μπορέσετε να με καταλάβετε και να καταλάβουν και οι υπόλοιποι απευθείας. Λοιπόν, η ΕΣΜΑ τακτικά τονίζει τους κινδύνους από το περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων. Υπάρχει η τάση από τους επενδυτές να ψάχνουν υψηλότερες αποδόσεις. Και αυτό που έχουμε δει είναι ότι ακριβώ επειδή γίνεται αυτή η προσπάθεια, τα funds ψάχνουν προϊόντα τα οποία δίνουν καλύτερες επιστροφές, εμοχλευμένα ή ψάχνουν εκεί που υπάρχει λιγότερη ρευστότητα. Οπότε το ερώτημα είναι ποιο είναι το αποτέλεσμα του περιβάλλοντος αυτού χαμηλών επιτοκίων που έχουμε τώρα περίπου εδώ και 10 χρόνια. Βλέπουμε ότι οι επενδύσεις αυτές αποτελούν πολύ μεγάλο μέρος του οικονομικού συστήματος. Τα χαμηλά επιτόκια και η προσπάθεια για ψηλέ αποδόσεις και το θέμα της ρευστότητα είναι καθοριστικά στοιχεία και όπως ξέρετε τα ταμεία τα επενδυτικά, τα usage, τα οσάκα δηλαδή, έχουν την υποχρέωση καθημερινά να ενημερώνουν τους επενδυτές τους και να γνωρίζουν αυτό το κίνδυνο. Το γνωρίζουμε και εμείς και γι' αυτό έχουμε φροντίσει να υπάρχουν μέσα και εργαλεία για λιγότερους κινδύνους. Να υπάρχει διαφάνεια, δημοσιεύουμε και έκθεση η οποία δείχνει ποια είναι η ρευστότητα του κάθε χαρτοφυλακίου και πόσο γρήγορα μπορούν να ζητήσουν τις επενδύσεις τους οι επενδυτές, πόσο γρήγορα μπορούν να πάρουν τα χρήματά τους πίσω δηλαδή. Αυτό που βλέπουμε τώρα σε εναλλακτικά ταμεία είναι ότι όντως οι μεγαλύτεροι κίνδυνοι βρίσκονται στον ε, τομέα της στέγασης. Πάντως η διαφάνεια είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτή είναι μια απάντηση που δίνουμε. Η άλλη είναι η κατάλληλη νομοθεσία από εσά και από το Συμβούλιο. Τα στρες τεστ, για παράδειγμα, οι δοκιμές αντοχής αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο για να εντοπίζονται οι κίνδυνοι ρευστότητας, κάτι το οποίο ε, έχει καταστεί υποχρέωση από τους διαχειριστές των επενδυτικών ταμείων. Σας είπα για το ΣΑΚΑ και για τις εναλλακτικέ επενδύσεις τι εφαρμόζουμε και επίσης χρησιμοποιούμε και κάποιες προσωμιώσεις δοκιμών αντοχής όπου εκεί ξέρουμε ότι μπορούν να τα καταφέρουν κάποια επενδυτικά ταμεία, αλλά υπάρχουν κάποια άλλα τα οποία είναι υψηλών αποδόσεων και που εμείς κρίνουμε ότι μπορεί εύκολα να έχουν δυσκολίες. Οπότε κάνουμε αυτές τις προσωμιώσεις. Τώρα κατά τα άλλα πρέπει πιο συγκεκριμένα να πω ότι οι εποπτικές αρχές φυσικά και παίζουν ένα σημαντικό ρόλο ε, σήμερα που έχουμε χαμηλές αποδόσεις και χαμηλά επιτόκια, αλλά να ξέρετε ότι δεν είναι κάτι το οποίο προκαλείται μόνο από τη νομισματική πολιτική. Σίγουρα η νομισματική πολιτική ε, απαντάει, προσπαθεί να απαντήσει σε διάφορα φαινόμενα, αλλά είναι και η γύραση του πληθυσμού, είναι και άλλοι παράγοντες οι οποίοι οδηγούν σε αυτό το περιβάλλον που γνωρίζουμε σήμερα. Ευχαριστούμε, κύριος Κουσμάου. Γκουε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, να σας το πω στα πορτογαλικά. Κύριε Κάμπα, εγώ θέλω να επανέλθω σε αυτό που, ο κύριος, είπαμε και ο κύριο Φάρκα, τον εκτελεστικό σας ε, διευθυντή. Το του είναι πολύ σημαντικά και ακριβώς με την ανάπτυξη της ε, θέσεως αυτής τώρα υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ε, έδωσε η EBA την ε, αδειά τη, το πράσινο φω για να γίνει αυτή η μεταγραφή. Υπάρχουν βέβαια οι προποθέσει που έχουν τεθεί, όμως κανείς πολίτη δεν μπορεί να θεωρήσει ότι αυτό ή αποτελεί μια εξασφάλιση από τους κινδύνους που δημιουργούνται από τις συγκρούσεις συμφερόντων. Οπότε, πρώτα-πρώτα έχουμε αυτό το θέμα της επαφής του λόγω κυρίου με το προσωπικό. Ε, φυσικά οκτώ χρόνια δουλεύει εκεί, οπότε έχει αναπτύξει κάποιες σχέσεις και τώρα ε, υπό την καινούργια του ιδιότητα μπορεί να έχει ε, και τηλεφωνικές επαφές ε, επίσης είπατε ως προϋπόθεση τι θα γίνει, πώς θα μπορέσουν οι, οι αρχές να δουν με τι θέματα θα ασχολείται στην καινούργια του δουλειά ο κύριος Φάρκας. Νομίζω ότι είναι αφελής αυτή η νέα ρύθμιση. Μα η νέα δουλειά του κυρίου αυτού άμεσα σχετίζεται με αυτό που έκανε στην υπηρεσία σας επί 8 ε, χρόνια. Οι αρχές δεν ανησυχούν και δεν θα πρέπει να εξασφαλιστεί ότι με ανεξάρτητο, με, με αμερόλητο τρόπο θα υπάρξει κάποιος έλεγχος. Γι' αυτό θέλω να μου πείτε. Πώς αποφασίσετε ό,τι αποφασίσατε και γιατί δεν κάνατε την ένσταση που δικαιούστε, δηλαδή να μην μπορέσει να λάβει καινούργια του θέση ο κύριος Φάρκας. Τέλος πάντων θα μπορούσατε να έχετε μια άλλη μεταβατική περίοδο μέχρι όταν λάβετε νέα του καθήκοντα. Κάμπα. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Σίγουρα και από την αρχή το σιγουρέψαμε ότι ε, από την αρχή υπάρχει θέμα με σύγκρουση συμφερόντων. Γιατί ήταν εκτελεστικός διευθυντής σε εμά. Το είπατε κι εσείς. Το ξέρουν. Όλοι αυτό το θέμα είναι πώς θα διαχειριστούμε το πρόβλημα. Εμείς ακολουθήσαμε το τι προβλέπει ο κανονισμός. Αυτό επιτάσσει ο νόμος. Δηλαδή, οποιοδήποτε από το προσωπικό, αφού αποχωρήσει, θα πρέπει να αναφέρει το τι δουλειά θα κάνει ε, τα επόμενα δύο χρόνια. Άρα, δεν μπορεί κανείς υπάλληλο να παραβεί την υποχρέωση. Επόμενο, σύμφωνα με του κανονισμού, δεν υπάρχει σύμφωνο μετά του 24 μήνε. Άρα, εμεί αυτό κάναμε και αυτό ήταν η αφετηρία μα, αυτή η ρύθμιση. Άρα, βάλαμε αυτή την προπόθεση για αυτά τους 24 ε, μήνες ε, και είπαμε ότι αυτό ξεκινάει 6 μήνες αφού λαμβάνει οποιαδήποτε απόφαση ε, χωρίς να έχει ήδη αναλάβει κάποια άλλη δουλειά. Άρα πρόκειται για ακόμα μεγαλύτερο διάστημα στην πράξη. Και έχουμε αυτού τους 18 μήνε που προστίθενται ε, στο εξάμεινο, άρα έχουμε 24 μήνε. συνολικά. Τώρα, όσον αφορά το πώ θα εφαρμοστεί αυτή η διάταξη, όντω. όπως είπαμε και στον κύριο Γαρικάνο, κάθε προϋπόθεση εφαρμόζεται σε διαφορετικό μέτρο. Είπαμε, κανείς υπάλληλος δεν ε, μπορεί να έρθει σε επαφή 18 μήνες αφού απεχώρησε ο κύριος ε, Φάρκα με αυτόν. Και όσον αφορά τους ε, τρίτους, ο κύριος Φάρκας έχει την ευθύνη να υλοποιήσει την ρύθμιση αυτή. Αν υπάρξουν ε, ενδείξεις, εμείς βέβαια θα ενεργήσουμε ανάλογα. Τώρα, όσον αφορά το αν μπορούσαμε ή όχι να το απογορεύσουμε να λάβει ε, αυτά τα νέα του καθήκοντα. Είναι δικαίωμά του όμως. Έτσι μας το είπε η νομική υπηρεσία. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε σε κάποιον κάτι τέτοιο. μπορούμε να προβούμε στου περιορισμού αυτού σε σύγκρουση συμφερόντων, αλλά όχι παραπάνω. Δεν μπορούμε να μην ε, κάνει αυτή την καινούργια δουλειά. Αν θέλει. Δεν υπάρχει διάταξη που να μπορεί να απαγορεύσει κάτι τέτοιο. Ε, τώρα σε σχέση με τους υπόλοιπους ε, υπαλλήλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εκτελεστικοί διευθυντές έχουν συγκεκριμένη θητεία και άπαξε κάποιο ε, αποχωρήσει, δεν προβλέπεται κάποια αποζημίωση. Επομένω, με το που φεύγει κάποιο από αυτή τη θέση, εκτελεχώ διευθυντή δηλαδή, έχει μηδέν ε, έσοδα, μηδέν εισόδημα. Αυτό αν κάνει κάποια άλλη δουλειά. Γι' αυτό και άλλα ισχύουν ε, σε σχέση με τους υπαλλήλους Ευρωπαϊκής Ένωση, σε σχέση με τη σύνταξή τους κλπ. Αυτά λάβουμε υπόψη για τη σχετική απόφαση. Σας ευχαριστώ. Τώρα για το ΕΛΚ, κύριο Μπέργκερ. Ε, ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ερώτηση προς τον ε, κύριο Κάμπα. Τον ε, προηγούμενο μήνα μας προειδοποιήσατε για το νόμισμα που προγραμματίζει Facebook το λεγόμενο Libra και μας είπατε πως Αυτά είναι αποκλειστική έκδοση κεντρικών τραπεζών και κρατών και προτείνεται έναν κανονισμό για κρυπτονομίσματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάτι με το οποίο μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε. Το ερώτημά μου είναι το εξή. Σε ποιο βαθμό οι εποκτικές αρχές είναι προετοιμασμένες ε, για να παρέμουν ρυθμιστικά σε τέτοια θέματα. Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι η Η ρύθμιση είναι η σωστή στρατηγική ή μήπως θα ήταν καλή ιδέα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να έκανε μόνη της ε, κάτι τέτοιο και να αναπτύξει ένα τέτοιο νόμισμα. Σας ευχαριστώ. Thank you. Thank you for the question. ευχαριστώ για την ερώτηση για τη Λίβρα και τα κρυπτονομίσματα. Πολύ σημαντικό θέμα και ερώτημα. Εκτός από μια σύσταση προς την Κομισιόν φέτος ε, τονίζοντας ότι στον τομέα των κρυπτονομισμάτων υπάρχει η πιθανότητα πολλά από τα στοιχεία και τα μέσα που υπάρχουν στην αγορά να μην μπορούν να ταυτοποιηθούν εύκολα με τον τρεχόντα κανονισμό που έχουμε δύο μεγάλες κατηγορίες. Ε, αυτά ας πούμε θεωρούνται ηλεκτρονικό χρήμα και εμπίπτουν στον κανονισμό περιπληρωμών είτε ως επενδυτικό προϊόν και θα εμπίπτουν στον σχετικό κανονισμό. Όμως κάποια από αυτά τα στοιχεία έχουν χαρακτηριστικά που δεν εμπίπτουν σε κάποια από αυτήν την κατηγορία. Και αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση της ε, Λίμπρα. Και βεβαίως αυτό αναφέρθηκε και στην σχετική έκθεση των ε, G7 για το πώς ακριβώς μπορούμε να καθορίσουμε την ε, δομή. Και βεβαίως αυτό υπήρχε στις ερωτήσεις που έστειλε η Κομισιόν ε, στην Ένωση των εκδοτών της Λίμπερα για να δούμε τι ακριβώς προϊόν είναι αυτό. Έχουμε λοιπόν αυτή την πρόκληση μπροστά μας. Πρέπει να είμαστε πιο σαφείς στο να αντιληφθούμε το τι είδους ε, ε, μέσα έχουμε για τα διάφορα προϊόντα. Και χάρηκα που ο Ντομπρόφσκης ανέλαβε την αξιολόγηση του υφιστάμενου ρυθμιστικού πλαισίου και να πούμε είτε είναι επενδυτικό προϊόν είτε ηλεκτρονικό χρήμα και να ρυθμιστεί αναλόγως. Αυτό λοιπόν, πέρα από άλλα ζητήματα όπως αναφέρατε, παραδείγματο χάνει την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής ή έκδοση από τις τράπεζες τέτοιων νομισμάτων που ξεφεύγουν από τον κανονισμό. Σας ευχαριστώ. Πολ Τάγκ, Σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ πολύ για τον κύριο Κάμπα. Είδατε την αντίδραση όχι μόνο εδώ αλλά και εκτός για τις περιστρεφόμενες θύρες. Το θέμα δεν είναι μόνο για τον Βάρκας ή για το EBA, είναι η εντύπωση που λέει ότι αν είσαι φιλικός προς τον κλάδο θα ανταμυφθείς με μια θέση στον κλάδο αργότερα. Αυτό είναι το πρόβλημα. προσπαθείτε τη σύγκρουση συμφερόντων να διαχειριστείτε όπως λέτε. Πόσο βέβαια αξιόπιστο μπορεί να είναι κάτι τέτοιο με πιστολή για αλλαγέ ότι ο κύριος Βάρκας δεν πρέπει να ασχολείται με θέματα όπως είναι η Βασιλεία 3 ή τα μη ξυπηρετούμενα δάνεια. Ναι, αλλά εγώ δεν βλέπω τι μπορεί να είναι αυτό που, με το οποίο θα ασχοληθεί και το οποίο δεν θα έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών. Πείτε μου εσείς ένα παράδειγμα. Και με όλα έχει ασχοληθεί ο κύριος Φάργας. Και έπειτα στην επιστολή λέτε ο κύριος Φάρκας είναι ο κύριος υπεύθυνο για να διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν οι προδιαγραφές. Δηλαδή εσείς επιβάλλετε κάποιες, κάποιους περιορισμούς και εκείνο θα ελέγχει το κατά πόσο τηρούνται αυτοί οι περιορισμοί ή όχι. Μα τι είναι αυτό, δεν υπάρχει καμιά αξιοπιστία σε αυτό. Ούτε μπορείτε να περιμένετε ότι ο κύριος Βάρκας δεν θα κάνει τίποτα, θα κάθεται στο γραφείο του και δεν θα ασχολείται με τα πιο σημαντικά θέματα και ούτε θα συνομιλεί με τους ομολόγους από την Ευρωπαϊκή ε, Τραπεζική Αρχή. Λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να εμποδίζονται πλήρως αυτές οι μετακινήσεις. Έπειτα, η αρχή μπορεί είτε να τον εμποδίσει να αναλάβει αυτά τα καθήκοντα ή και μετά το υπόλοιπο. Λοιπόν, η κατάσταση προσωπικού σας επιτρέπει να εμποδίσετε αυτήν τη μετακίνηση. Οπότε γιατί δεν το κάνετε. Κατά τα άλλα, για να γραφτεί στα πρακτικά, εκτίμησα την απάντηση του κύριο Καργκάνο, νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν πρέπει να έχουν καμία επαφή με τον κύριο Φάρκα. Δεν πρέπει να επιστρέψουμε κάτι τέτοιο. Είναι πολύ βασικό για την ακαιρεότητα του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ο κύριο Κάμπα. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να διευκρινίσουμε, οπότε χαίρομαι που έχει δημοσιοποιηθεί τόσο πολύ. Και επανέρχομαι στην ερώτησή σας. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι ούτε υπέρ του κύριου ούτε της ε, ΕΣΜΑ να υπάρχει συμπεριφορά που θα εκλαμβάνεται σαν παραβίαση της απόφασης που λάβαμε. Τα είπα και στον κύριο Καρικάνο. Εγώ δεν περιμένω ότι θα έρθει ο κύριος Φάρκας. Αλλά αν έρθει, είναι σημαντικό να μας ενημερώνετε αν υπάρχει παραβίαση. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Ο καλύτερος τρόπος. Τώρα, όσον αφορά το αν μπορούμε να εμποδίσουμε την απόφαση. Και έρχομαι στην απάντηση που έδωσε και στην προηγούμενη ερώτηση. Είναι σημαντικό και αυτή ήταν η νομική συμβουλή που πήραμε. Είναι ότι πρέπει να ζυγίζουμε την κατάσταση. Και εδώ εμποδίζουμε κάποιον να έχει τη δυνατότητα να κερδίσει τη ζωή του χωρίς να του προσφέρουμε μια εναλλακτική λύση. Περί αυτού πρόκειται. Γιατί όταν ο εκτελεστικός διευθυντής φεύγει από το ΕΠΑ. Εντάξει, μπορεί να έχει άλλες δυνατότητες, αλλά αυτή τη στιγμή αυτήν έχει. Οπότε η νομική απόφαση, η γνωμοδότηση που πήραμε ήταν να περιοριστεί το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων που θα αναλάβει στα νέα του καθήκοντα για να μην υπάρχει αυτή η σύγκρουση συμφερόντων. Αυτό τι σημαίνει, όπως είπατε. Σημαίνει ότι στα νέα του καθήκοντα ο κύριος Βάρκας θα πρέπει να ασχοληθεί με πράγματα τα οποία δεν συγκρούονται με τη σύγκρουση εφερόντων δηλαδή, με αυτά με τα οποία ασχολιόταν προηγουμένως. Υπάρχει εσωτερική οργάνωση, υπάρχει η αξιολόγηση κινδύνου ε, βάσει της εξέλιξης του κλάδου, υπάρχουν άλλα θέματα που είναι εκτός Ευρώπης θα μπορούσε να ασχοληθεί με τέτοια. Αλλά δεν θα το αποφασίσουμε εμείς αυτό. Για την επιβολή της απόφασης, προφανώς, σε αυτόν απευθύνεται η απόφαση. Και ο πρώτος που πρέπει να συμμορφωθεί, που είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί, είναι αυτός τον οποίο απευθύνεται η απόφαση. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να ε, συμμορφωθώ ε, με τον οδικό κώδικα κυκλοφορίας. Οπότε οι αρχές επιβάλλουν στο συγκεκριμένο άτομο στο οποίο απευθύνουν την απόφασή τους. Είναι κάτι προφανές, δεν είναι τίποτα περίεργο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε λοιπόν για το ρινιό τώρα. Σας ευχαριστώ και έχω τρει ε, ερωτήσεις και προ του τρει καλεσμένου. προς το τον σε σχέση με τη μετάβαση στην πράσινη εποχή και τη χρηματοδότηση. Εσείς είστε ικανοποιημένοι ότι για τις κεφαλαιογορές ε, αυτά τα, τα πράσινα ομόλογα πρόκειται να αρκέσουν στις αγορές και στους επενδυτές. Ε, για πέστε μας, αυτή η διπλή δημοτική πολιτική ε, θεωρείται ότι είναι επαρκής σε Ιρλανδία, στο Έμενο Βασίλειο και αλλού υπάρχει θέμα, οπότε θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με αυτή την διπλή ε, τιμολόγηση στην ε, ασφαλιστική αγορά. Κύριε έχουμε αυτά τα των δάνεια και έχουμε και τις ε, τράπεζες που θέλουν κάπως να ρυθμίσουν το πρόβλημα σε σχέση με τη συμφωνία της Βασιλείας 3. Πώς στηρίζονται και τα εθνικές αρχές ώστε να μην πηγαίνουν ε, σε κάποιες εταιρείες ε, αρπακτικών αυτά τα κόκκινα δάνεια και αυτοί μετά να λιμένονται τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις γιατί νομίζω ότι έχουμε χάσει το τρένο σε αυτό το μέτωπο. Θα πρέπει κάτι να γίνει με τις τράπεζες γιατί το πρόβλημα είναι οι κεφαλιακές απαιτήσει των τραπεζών που θέλουν να απαλλαγούν από τα κόκκινα δάνεια. Υπάρχει προστασία γιατί πολλές φορές κάποιος θα πρέπει να προστατεύει και τους καταναλωτές, τους περάτες των τραπεζών και ταυτόχρονα να είναι εποπτική αρχή για μια τράπεζα. Κύριε Μαγιώ, σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις. Το σημαντικό είναι το εξής όσον αφορά τα πράσινα ομόλογα, ότι εδώ σαφώς υπάρχει ζήτηση να ξεκαθαριστούν τα πράγματα, να υπάρχει περισσότερη αξιοπιστία όσον αφορά ε, το τι ορίζεται πράσινο ομόλογο. Ο φυσικά έχει προχωρήσει περισσότερο από το κρατικό για τα στάνταρ που θα ισχύσουν όσον αφορά αυτά τα ομόλογα και ακριβώς λόγω του κινδύνου του να υπάρχει ε, παράκαμψη νομοθεσίας, να υπάρχουν διαφορετικά στάνταρ, να υπάρχουν ε, διαφορετικές ρυθμίσεις, θα πρέπει να ξεκαθαριστεί το τοπίο όντως είναι σε εξέλιξη ο προβληματισμός για το ποιο θα είναι το πιο εύστοχο πλαίσιο κατά την προσωπική μου γνώμη. Τώρα ήρθε η ώρα να μπορέσουμε να έχουμε νομοθεσία, οπότε ε, να καθορίζεται το τι θα κάνει ο δημόσιος τομέας που τελικά θα πρέπει να αποφασίσει το τι συνιστά πράσινο ομόλογο επίσης στην πράξη κανείς θα πρέπει να μπορεί να ελέγξει κατά πόσον τα μόρια που κυκλοφορούν ανταποκρίνονται στις τεθήσεις προϋποθέσεις. Και ξέρουμε και από άλλους τομείς της οικονομίας ότι μπορεί να υπάρξει διασταύρωση από τους ε, τρίτους επαλήθευση δηλαδή. Αλλά είναι σημαντικό αυτή η τρίτη να μπορούν να θεωρήσουν ότι υπάρχει αξιοπιστία. Το ίδιο αφορά και με την υποβολή των εκθέσεων. Καταλήξαμε σε ένα σύστημα που διέπει το δημόσιο τομέα αλλά και οι, ίδιες, οι ίδιοι οι οικονομικοί ελεγκτές υπάγονται και υπόκειται σε αυτούς τους κανόνες. Άρα θα πρέπει και για τα πράσινομόλογα έτσι να προχωρήσουμε. Ε, Μπερναρντίνο, ευχαριστούμε για την ερώτηση. Θα πρέπει να δούμε τα πράγματα από πλευρά εποπτεία των επιχειρήσεων και έχουμε σχετικές εκθέσεις αιτήσει και βλέπουμε ποια είναι τα βασικά ζητήματα από κάθε κράτος μέλος. Και όχι μόνο από τις υποπτικές ε, αρχές, αλλά από του καταναλωτές, από την αγορά και έτσι καθορίζουμε ποιες είναι οι προτεραιότητε και σε ποια μέτωπα. Ας πούμε έχουμε αυτή την θεματική ε, αξιολόγηση για ταξιδιωτική ασφάλιση, είχαμε προβλήματα σε μια σειρά κρατών, ακριβώς από πλευράς ε, τιμολόγηση επιτροπών ε, συγγνώμη, προμηθειών και εμεί κινηθήκαμε αναλόγως. Η διπλή τιμολόγηση είναι όντω ένα θέμα, όπως είπατε, σε Αγγλία Ιρλανδία και αυτό οπωσδήποτε θα είναι η προτεραιότητά μας στο άμεσο μέλλον. Δεν αποκλείω το να προβούμε σε μια ανάλυση πανευρωπαϊκή. Αλλά υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως είπαμε, δηλαδή η σύνδεση ασφαλιών με στεγαστικά, να υπάρχει διαφάνεια η σύνδεση ασφαλιστικών συμβολέων με άλλα προϊόντα. Όλο ένα και πιο πολύ επεκτείνεται στην Ευρώπη αυτή η πρακτική. Άρα να γίνει αυτό προτεραιότητα, να κάνουμε πανευρωπαϊκή ανάλυση. Σίγουρα, σίγουρα αυτό το οποίο είπατε για την πλήρη το προσέχουμε και είμαστε σε επαφή σε σχέση με αυτό με τι εθνικέ αρχέ. Κάμπα. Σα ευχαριστώ για το ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων ε, δανείων. Γνωρίζετε ότι δεν ισχύει το ίδιο σε όλες τις ε, χώρες. Ε, κάποιες χώρες έχουν υψηλό επίπεδο με εξυπηρετούμενων δανείων και ο ρυθμός της ε, μείωσης εξαρτάται. Κάποιες φορές το αναλαμβάνει μια εταιρεία, άλλες φορές γίνεται από το κράτος και υπάρχει αρκετά μεγάλη μετάδοση των μη εξυπηρετούμενων δανείων εκτός της οικονομίας και των ε, τραπεζών. Οπότε έχουμε διαφορετικές ε, προσεγγίσεις και πάρα πολύ μεγάλες ε, διαφορές για να είμαι ειλικρινής. Το θέμα το οποίο αναφέρατε τώρα συγκεκριμένα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα άτομα είναι θέμα προστασίας των πελατών, δηλαδή αν αυτά τα κάνουν οι τράπεζες, κάτι το οποίο επίσης διαφέρει ανά την Ένωση. Τι αφορά ακριβώς και κάποιες χώρες που έχουμε δύο που έχουν μεγάλη δυσκολία εκτέλεσης ενός ε, μη εξπερτωμένου δανείου ε, εις βάρος ενός ε, οφειλέτη. Δηλαδή είναι δύσκολο να βρούμε λεπτομερείς πληροφορίες. Θα εκδώσουμε την έκθεση μας για την εκτέλεση των μη εξυπηρετούμενων δανείων Οπότε θα επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες, αλλά βεβαίω αυτό ακολουθεί μόνο την εκτέλεση δανείων που δίνουν οι τράπεζες ε, σε κάποιο τρίτο μέρος που δεν είναι τράπεζα και τις εκτέλεση Σε αυτή την περίπτωση βεβαίως αν δεν είναι τράπεζα δεν έχουμε κάποια αρμοδιότητα. Αλλά θα έχουμε περισσότερες ε, πληροφορίες και ευχαριστώ ε, να σας δώσουμε. Έχουμε, τώρα έχουμε λοιπόν 10 λεπτά και πέντε άτομα που έχουν να κάνουν ερωτήσεις. Οπότε σας παρακαλώ να είστε σύντομοι. ορί για το όλοι. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω την ε, μητρική μου γλώσσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δύο ερωτήσεις έχω προς τον κύριο Κάμπα και θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Η πρώτη μου ερώτηση είναι η εξής εξετάσαμε την οικονομία τα τελευταία χρόνια. Υπήρχε ανάπτυξη, η ανεργία μειωνόταν, οι τράπεζες τα πήγαιναν μια χαρά. Ταυτόχρονα όμως βλέπουμε ότι η εμπιστοσύνη των ανθρώπων στον κλάδο δεν είναι η μεγαλύτερη και ο κόσμος φοβάται ότι υπάρχουν ε, λιγότερες τράπεζες που κόπηκαν στα τρες τεστ από ό,τι θα έπρεπε. Και ο Σεν λέει τα σχετικά έγγραφα στην Επιτροπή ε, τη δική μας ε, και είχαμε πληροφορίες για την Deutsche Bank και η εμπορική αξία της, της οποίας είναι πολύ καλύτερη από την ονομαστική της αξία. Και θα ήθελα να γνωρίζω γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δεν πιστεύει ο κόσμος ότι οι τράπεζες ε, τα πάνε μια χαρά. Η δεύτερη ερώτηση αφορά τα κρυπτονομίσματα. και θα ήθελα να αφαιρθώ στην ε, ρύθμιση και την προσέγγιση των ε, τραπεζών. Αυτό είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος γιατί οι τράπεζες κάνουν χιλιάδες ε, πελάτες. Εγώ προσφάτως ήθελα να πληρώσω σε μια τράπεζα και μου είπαν «Α, όχι δεν γίνεται μόνο με Revolut. Πραγματικά σοκαρίστηκα. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς τις τράπεζες ως Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή πώς ε, θα επιζήσουν. Έχουμε προβλήματα ξεπλήματος χρήματος, τρομοκρατίας και άλλες δυσκολίες, αλλά και τα κρυπτονομίσματα ήταν δυσκολία. Πώς θα επιβιώσουν οι τράπεζες το ότι χάνουν τους ε, πελάτες τους. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Έχετε απόλυτο δίκιο όταν λέτε ότι η αντίληψη των επενδυτών ε, της αγοράς για τις ευρωπαϊκές ε, τράπεζες ε, ε, δεν είναι θετική και η αξία αγοράς σε σχέση με την ονομαστική αξία είναι χαμηλότερη και βεβαίως το ερώτημα είναι το γιατί προσπάθησα να εκθέσω κάποιους λόγους, κυρίως το μακροπεριβάλλον χαμηλών επιτοχίων, η χαμηλή ανάπτυξη σε πολλές χώρες της Ένωσης, ε, Βεβαίω σημαντική πτυχή, η αδυναμία των τραπεζών να προσαρμόσουν τα έσοδά τους στο κόστος, οπότε η αναλογία κόστους εσόδων δεν αυξάνεται. Και επίσης είπατε και εσείς ε, στο δεύτερο ερώτημά σας η πρόκληση από την τεχνολογία και τα νέα εναλλακτικά προϊόντα είναι πάρα πολύ μεγάλη για τον τραπεζικό τομέα σε σχέση με τις επενδύσεις που πρέπει να κάνουν για να ανταποκριθούν στις τεχνολογικές προκλήσεις και βεβαίως έχουμε και νέες εταιρείε που μπαίνουν ε, σε κομμάτι της δουλειάς τους. Παραδείγματος χάρη η Revolut που αφορά τις ε, πληρωμές ε, ε, σε άλλα νομίσματα, κάτι το οποίο παραδοσιακά έκαναν οι τράπεζε Είναι λοιπόν εδώ πέρα πω ο ανταγωνισμό έχει μειώσει το περιθώριο κέρδους, οπότε οι προκλήσει για τις τράπεζες είναι μεγάλε. Τι κάνουμε λοιπόν, ως ρυθμιστικέ αρχές ανησυχούμε, ε, έτσι ώστε, γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένα βιώσιμο μοντέλο για τις τράπεζες μέσω μακροπρόθεσμα και τα stress test έχουν δείξει ότι οι τράπεζες ε, είναι πιο ισχυρές, έχουν περισσότερο κεφάλαιο, λιγότερα εξυπηρετούμενα δάνεια και τα σχετικά άλλα. Όσον αφορά την ε, κερδοφορία, βεβαίως ε, αυτό το κομμάτι δείχνει σημαντικές αδυναμίες. Οι τράπεζες πρέπει να βρουν μια λύση. Το κόστος είναι ένα θέμα. Και βεβαίως θα πρέπει να α, επιβιώσουν οι ικανότεροι και οι υπόλοιποι να μόνο από την αγορά. Είναι σημαντικό αυτό. Και μια άλλη πτυχή είναι ότι εμείς ως ρυθμιστές πρέπει να γνωρίζουμε ότι από εδώ και μπρο ε, στην διαδικασία της τεχνολογικής κοινοτομίας θα πρέπει να είμαστε τεχνολογικά ουδέτεροι ως προς την τεχνολογία που εφαρμόζεται, αρκεί βεβαίω να πληρούνται κάποια κριτήρια προστασίας ε, των πελατών, ε, να διασφαλίζεται η χρηματοπιστωτική σταθερότητα, αλλά πρέπει να είμαστε ουδέτεροι και μεταξύ παικτών, μεταξύ εταιριών. Δηλαδή να μην προστατεύουμε, να προστατεύουμε τις τράπεζες σε σχέση με τις εταιρείες που δεν είναι τράπεζες. Το βασικό είναι να παρέχονται υπηρεσίες, όχι να προστατεύουμε τις τράπεζες ή κάποιες τράπεζες, μικρές, μεγάλες και τα σχετικά. Και αυτή είναι η πρόκληση η βασική που αντιμετωπίζουμε. Σας ευχαριστώ. Πέτρο Μάρκες σοσιαλδημοκράτες. Ευχαριστώ στον κύριο Μπερναρντίνο και θα μιλήσω πορτογαλικά. Πρόεδρε, για... επειδή είσαστε και πρόεδρος της ΕΙΟΠΑ, για αυτές τις αρμοδιότητες σας θέλω να μιλήσω. Η κατάσταση χαμηλών επιτοκίων είναι παράγοντας κινδύνου, όπως είπατε και στην αρχή για ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αλλά όταν μιλάμε για ασφάλειες και συντάξεις, τι συγκεκριμένα μέτρα μπορείτε να πάρετε για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα του κλάδου μέσα σε αυτό το πλαίσιο χαμηλού κινδύνου μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται τώρα. Τώρα, ως πρόεδρος της Μικτής Επιτροπής για την εποπτεία και για τους συστημικούς κινδύνους. Πώς εκτιμάτε την κατάσταση του χρηματοπιστωτικού τομέα στο σύνολό του. Γιατί μιλάμε για χαμηλό αλλά από την άλλη μεριά υπάρχουν πολλά στοιχεία που λείπουν για να συμπληρώσουμε την Κεφαλιακή Ένωση. Οπότε ρωτάω για σας, ποια θα ήταν η προτεραιότητα από πλευράς του δικού σας οργανισμού. Έπειτα, το σκιώδες τραπεζικό σύστημα. Μιλήσαμε πολύ για αυτό το θέμα. Είναι κάτι που έχει αυξηθεί πολύ ως φαινόμενο τα τελευταία χρόνια. Και η ερώτησή μου είναι, ρυθμίζουμε με το σωστό τρόπο αυτές τις δραστηριότητες του σκιώδους τραπεζικού συστήματος ή θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα. Απάντηση. Ευχαριστώ πολύ θα προσπαθήσω να σας απαντήσω στα αγγλικά για την πρώτη σας ερώτηση όσον αφορά για τον αντίκτυπο του περιβάλλοντος χαμηλών επιτοκίων που διαρκεί και μάλιστα αρνητικών επιτοκίων μερικές φορές. Ε, φυσικά και είναι μια ανησυχία για τις συντάξεις και τις ασφαλίσεις, γιατί το επιχειρηματικό μοντέλο που προβλέπετε μέχρι τώρα τίθεται υπό αμφισβήτηση. Και εμείς βέβαια λαμβάνουμε ήδη μέτρα εδώ και χρόνια. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι έχουμε ένα καθεστώς με την οδηγία Φερεγγιότητα 2 που προλαμβάνει και παρακολουθεί την αξιολόγηση της αγοράς και προσφέρει τόσο στους επόπτες όσο και στην αγορά ε, καλύτερη κατανόηση για τις επιπτώσεις των αλλαγών και κυρίως των χαμηλών επιτοκίων. Τώρα με την φερικιότητα 2 έχουμε ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται ε, καλύτερα, πιο κοντά παρακολουθεί τις προκλήσεις των χαμηλών επιτοκίων. Και αυτό είναι πολύ θετικό. Και φαίνεται και από τα μέτρα τα οποία έχει πάρει η ΕΙΟΠ ήδη και μερικά χρόνια, ώστε να προσαρμοστεί το επιχειρηματικό μοντέλο ακριβώς των επιχειρήσεων και το κάνουν, προσαρμόσουν καλύτερα τις εγγυήσει που βάζουν στην αγορά. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι πολύ σημαντικά, αλλά επίσης πολύ σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι χειρίζεσαι καλά τα ήδη υπάρχοντα χαρτοφυλάκια, γιατί είναι αυτά ακριβώς που προβλέπουν τις υποχρεώσεις απέναντι στους Ευρωπαίους καταναλωτές. Και με την φερικιότητα 2 φροντίσαμε να υπάρχει μια μεταβατική μεν περίοδος, αλλά όχι ανοιχτή στο δινεκές και μέσα σε αυτό το διάστημα θα έπρεπε οι επιχειρήσεις να ανεβάσουν τα κεφαλαιακά τους αποθέματα. Επίσης, οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να διασφαλίσουν ότι η πολιτική τους μερισμάτων λαμβάνει υπόψη την αναγκαιότητα ε, αύξησης του κεφαλαίου ε, με τα χρόνια. Οπότε και αυτό είναι πολύ σημαντικό και το παρακολουθούμε συνεχώς. Τώρα τι μπορεί να γίνει παραπάνω. Δύο πράγματα. Όσον αφορά τις δοκιμές αντοχής πρώτα. Και πρέπει να πω ότι εδώ και δύο χρόνια κάνουμε τέτοιες δοκιμές της ασφαλίσεις και της συντάξεις και πολλές φορές μας έχει επικρίνει ο κλάδος ότι κάνουμε υποθέσεις που δεν ήταν καθόλου ρεαλιστικές, ας πούμε, για τα επιτόκια. Ενώ αποδείχθηκε ότι είχαμε δίκιο, γιατί πριν από χρόνια είχαμε κάνει μια τέτοια δοκιμή αντοχής με σενάριο χαμηλών επιτοκίων και σας πληροφορώ ότι η πραγματικότητα μας ξεπέρασε πολύ γρήγορα. Οπότε είναι σωστό και από πλευράς εποπτείας και από πλευράς επιχειρήσεων να προλαμβάνουν ε, τις καταστάσεις και να φροντίσουν να είναι βιώσιμες οι επιχειρήσεις τους. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο για το οποίο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί η σημερινή κατάσταση χαμηλών επιτοκίων φέρνει όπως είπα, και αλλαγές στο επιχειρηματικό μοντέλο, αλλά και στις εγγυήσει που δίνονται. Και περνάμε τώρα σε ένα περιβάλλον ε, μεταφοράς και αυτό με τη δικιά του την ε, σειρά οδηγεί σε άλλα ζητήματα. Οι επιχειρήσεις έχουν επιλογές για τις ε, επενδύσει που κάνουν, χωρίς όμως να ξέρουν πάντα με τι κριτήρια να το κάνουν και πώς να το κάνουν αυτό. Τώρα πρέπει να παρακολουθούμε καλύτερα αυτά τα προϊόντα, αυτά τα ασφαλιστήρια, ώστε με τα χαμηλά επιτόκια ο κίνδυνος να μην μεταφέρεται στον καταναλωτή για το συστημικό κίνδυνο. Τώρα μπορώ να σας δώσω την προσωπική μου άποψη. Σαφώς και πρέπει να ολοκληρωθεί η κεφαλαιακή ένωση. Όταν έχουμε ευρωπαϊκά προϊόντα, η εποπτεία πρέπει να είναι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με τα ΠΕΠΣ e δεν ήταν εφικτό αυτό, δεν ήταν δυνατόν. Αυτή ήταν η πρόταση της Επιτροπής. Το Κοινοβούλιο μας στήριξε, αλλά δεν συμφώνησε το Συμβούλιο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να συζητηθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο περισσότερο. Σκοτ και του ευχαριστώ. Για τον κύριο Μάγερ θέλω να ρωτήσω. Αυτό το θέμα της βιωσιμότητας της κεφαλαίου αγοράς. Τον Ιούλιο του 19 εκδώσετε κάποιες συμβουλές όσον αφορά ε, τις εταιρείες αξιολόγησης. Δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί ο κανονισμό CRA ούτως ώστε να μπορέσει να ανταποκρίνεται με αυτά ε, που θεωρούμε ότι είναι βιώσιμα γιατί αυτές οι εταιρείε αξιολόγηση ε, για τις κεφαλαιακές ροές είναι πάρα πολύ σημαντικέ Στον Ιούνιο του 2018 είπαμε ότι η ΕΣΜΑ θα πρέπει να έχει την εντολή να απαιτεί από αυτέ τι εταιρείε να έχουν τη μεθοδολογία του και την αξιολόγηση για κίνδυνο. Οπότε εάν ε, δεν το κάνετε αυτό τότε τι, βλέπετε ως βιώσιμο προς τους επενδυτές σε σχέση με τις εταιρείε αξιολόγησης και πώς θα μπορέσετε να κατευθύνετε τις επενδύσεις εκεί που θέλουμε για την προσπάθειά μας για αντιμετώπιση αλλαγής του κλίματος. Επίσης, κεφαλογίες πώς νομίζετε ότι θα προετοιμαστούν για, τις, ε, για τα οικονομικά σοκ σας ευχαριστώ για την ερώτηση και να αρχίσουμε από το τέλος. Ότι θα πρέπει να δούμε τα θέματα βιωσιμότητας από πλευράς των κεφαλαιογορών και έτσι να εξασφαλίσουμε το ότι θα πρέπει να υπάρχουν προφορές για κάποιες εταιρείες ε, όσον αφορά το περιβάλλον, ε, να, υπάρχουν σχετική, να υπάρχει σχετική ενημέρωση, αλλά και αυτό να λαμβάνει υπόψη και στην αξιολόγηση των εταιριών αυτών και το είπαμε και φέτος ότι είχαμε τον παράγοντα βιωσιμότητα, το οποίο μετρούσε για την αξιολόγηση. Αυτό θα πρέπει να ξεκαθαριστεί, αυτό θα πρέπει να το ξέρουν οι επενδυτές, αλλά θα πρέπει να πούμε και το ότι ε, κάθε αξιολόγηση θα πρέπει να περνάει μέσα από τη βιωσιμότητα, γιατί είχαμε κάποιες ε, εταιρείες όπου αυτό δεν ελαμβάνεται υπόψη στην αξιολόγηση επίση. Δεν είναι μόνο το θέμα του περιβάλλοντος, είναι και το τι κάνει η εταιρεία, τι κάνουν οι επενδυτές που θέλουν πληροφορίες, γιατί πέραν της αξιολόγησης της δυνατότητας αποδόσεων θα πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι οι επιπτώσεις για το περιβάλλον. Οπότε είναι αυτό σημαντικό να ληφθεί υπόψη. Εμείς αυτό θέλουμε και το είπαμε ε, και αρχάς του είπαμε στην Κομισιόν για το πώς θα πρέπει τα ταμεία και οι επενδυτικές εταιρείε να λάβουν υπόψη επιπτώσεις στο περιβάλλον όποτε συμβουλεύουν πελάτες είπαμε ότι δεν θα είναι έξυπνο κανείς να ασχοληθεί μόνο με την φερεγγιότητα όσον αφορά την αξιολόγηση, αλλά θα πρέπει η αξιολόγηση πέραν της εφερεγγιότητας αλλά υπόψη και το περιβάλλον, γιατί οι αξιολογήσεις αυτών των φορέων σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό αφορούν την αξιολόγηση του αξιόπιστου. Και πολλές φορές αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Γκούναρ Σας ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Έχω μία ερώτηση για τον κύριο Κάμπα και θα μιλήσω γερμανικά τα τελευταία τρία χρόνια το 5% των ασθενέστερων τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σύμφωνα με τον πίνακα βαθμολογίας ε, της EBA εδώ από το δεύτερο τρίμηνο του 2019 δεν έχουν αυξήσει την ε, ικανότητα επιβίωσής τους. Λοιπόν, τρεις ερωτήσεις έχω. Πρώτον, Κατά την άποψή σας, ε, τα στατιστικά αυτά στοιχεία αποδεικνύουν ότι οι απαιτήσει ε, κεφαλιακές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα μέτρα μείωση του κινδύνου έχουν αποτύχει, καθώς ε, δεν έχει αυξηθεί η επιβιωσιμότητα των τραπεζών και έτσι οι μεγαλύτερες τράπεζες παραμένουν συστημικός κίνδυνος παρά την Βασιλεία και τις σχετικές διατάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ίδια κεφάλαια. Δεύτερον, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις πολλών γερμανικών τραπεζών, τα αρνητικά επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η έκδοση χρήματος έχουν επηρεάσει την βιωσιμότητα των τραπεζών. Εσείς πώς εκτιμάτε την ε, πλημμυρίδα χρήματος ε, της ΕΚΤ όσον αφορά την ε, επιβίωση των τραπεζών. Και τέλος, τα αρνητικά επιτάκια οδηγούν σε άμεσο κόστος της τράπεζας και σε έμεσο κόστος μέσω του margin squeeze. Ιδιαιτέρως σε χώρες στις οποίες είναι παράνομο να χρεώνουν αρνητικά επιτόκια στους καταθέτες. Θα υπάρξει λοιπόν κάποια χαλάρωση για να βελτιωθεί η ικανότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα να ανταποκριθεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Κάμπα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσον αφορά την πρώτη πτυχή, όπως είπα στις αρχικές μου παρατηρήσεις, η κεφαλαιοποίηση και τα σχετικά ποσά των ευρωπαϊκών τραπεζών έχουν βελτιωθεί. Αλλά έχει μειωθεί η διασπορά, δηλαδή οι τράπεζες αυτές με τα μικρότερα ποσοστά κεφαλαιοποίησης. Οπότε θεωρούμε ότι έχει υπάρξει σημαντική προσπάθεια και τα κεφάλαια αυτή τη στιγμή είναι λίγο πολύ σύμφωνα με τους ε, κανόνες και σύμφωνα με τα stress test όπως είπαμε δεν υπάρχουν πλέον ανάγκες ουσιαστικές ε, κεφαλαιοποίησεις. Βεβαίω αυτό το οποίο έχει σημασία είναι η προοπτική κερδοφορία η οποία δεν είναι πολλά υποσχόμενη και έχουμε και τα χαμηλά επιτόκια που είναι βεβαίως, κάνουν την κατάσταση δύσκολη για το εισόδημα των τραπεζών και ταυτόχρονα οι τράπεζες έχουν δείξει δυσκολίες στο να ανταποκριθούν στο θέμα του κόστους βεβαίως το θέμα των εσόδων να αντισταθμίζεται από ένα πολύ ευνοϊκό περιβάλλον το οποίο καταλήγει σε χαμηλότερες ε, ε, προβλέψεις ε, γιατί βεβαίως αν η οικονομία παρουσιάσει ύφεση θα μπορούσαν να ασκηθούν ακόμη μεγαλύτερες πιέσεις στις τράπεζες. Για το τρίτο θέμα το οποίο αναφέρατε για το πώς θα μεταφερθούν αυτά στον ισολογισμό των τραπεζών και βέβαια το θέμα του πώς επηρεάζονται οι καταθέσεις και τα υπόλοιπα στοιχεία του ενεργητικού. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια αξιολόγηση στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή για το τι γίνεται, γιατί όπως ξέρετε αυτό διαφέρει από χώρα σε χώρα και μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για τις τράπεζες στο μέλλον ή ίσως και όχι. Αλλά θα μπορούσαν να αντιδράσουν σε άλλου τομείς αυξάνοντα παραδείγματο χάρη τι χρεώσει χρεώσεις ε, για τις διάφορες υπηρεσίες. Ε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Okay, thank you. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μπερναντίνο, τον κύριο Πάγκα και τον κύριο Μαγιόρ για τις απαντήσεις του στις ερωτήσεις μας. Ευχαριστώ και τους ευρωβουλευτές για τη συμμετοχή τους σε αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση. Προσβλέπουμε και εμείς σε παρετέρω συνεργασία. Ο κύριος ε, Γκούσμα θα αναλάβει τώρα. Dankeschön. Ja, ja, ja, ja mit äh, Frau Brock. You Thank you. Uh, we will now go on for... Πρόεδρος, πάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 7 και στο σημείο υπαριθμών 8 της ημερησίας διατάξεως. Παρακαλώ εσείς που βγαίνετε από την αίθουσα, κάντε λίγο πιο γρήγορα και οι υπόλοιποι καθίστε. So Lydia is the rapporteur for Έχουμε τώρα την την εισηγήτρια και των δύο αυτών σημείων των δύο εκθέσεων, την κυρία Περέρη που και ο κύριος Φέρμπερ θα την αντικαταστήσει. Ευχαριστώ συνάδελφοι να σα ε, διαβάσω ένα ενημερωτικό σημείο. Η ψηφιοποίηση αράζει τι ε, κοινωνίε μα και τι οικονομίε μα και οι καταναλωτές και οι εταιρείε. Ε, κάθε μέρα ε, υφίστανται ένα σοκ σε όλα τα μέτρα, σε όλες τις υπηρεσίες. Το ηλεκτρονικό εμπόριο αναπτύσσεται παγκόσμια και συγκεκριμένα στην Ευρώπη. Το 2018 είχαμε 69% των χρηστών του διαδικτύου που αγόραζαν το ίντερνετ και 68% από κάποιους που πολλούσαν κάτι σε άλλη χώρα. Και γι' αυτό θα πρέπει τώρα να δούμε την νέα ψηφιακή αγορά ως θέμα προτεραιότητας και μεγάλης ευκαιρίας τόνωση της οικονομίας. Ε, για αυτό θα πρέπει να έχουμε ευφύ νομοθεσία, μια νομοθεσία που θα ρυθμίζει αλλά δεν βάζει φραγμό στον ανταγωνισμό ε, και σε ένα ελεύθερο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις, καινοτομία και ψηφιοποίηση ε, χέρι-χέρι προχωρούν στις αγορές και η πληροφορική δεν θα πρέπει να είναι φραγμός, οπότε εγώ θέλουμε με αυτή την έκθεση να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στρατηγική για μοιρασμό της πληροφορίας και συνεργασία. Δυστυχώς. Λέει, δεν μπορούσα να έρθω όπως ήθελα σήμερα και ζήτησα από τη γραμματεία να μεταθέσει την συνάντηση για αύριο. Αλλά δεν κατέστη αυτό δυνατόν και συμπαθάτε με που αποσίασα αλλά περιμένω πώς και πώς να συνεργαστούμε για αυτές τις εκθέσεις και να ε, με συγχωρήσουν και οι σκιώδεις με τους οποίους θα εργαστούν τις επόμενες μέρες. Πιέζει το χρονοδιάγραμμα, ε, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε και θα έχουμε μια κοινή θέση του Κοινοβουλίου τελικά. Όπως γνωρίζετε πρόκειται για μια διαδικασία διαβούλευση για τις δύο εκθέσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι το Συμβούλιο ε, διαμορφώνει συνένεση, αλλά θα πρέπει να αναδείξουμε το ότι το Κοινοβούλιο έχει ξεκάθαρη θέση όσον αφορά την καταπολέμηση της απάτης περί των ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο και μες ρυθμίσεις ε, ε, γιατί πρόκειται για την καινοτομία και έτσι θα πρέπει να ενεργήσουν οι νομοθέτες. Σημαντικό το θέμα, ε, να έχουμε απλουστευμένη διαδικασία και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να τοποθετηθούν όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Θέλουμε τη συμβολή τους και έτσι να μπορέσουμε το θέμα αυτό να ενταχθεί στην ημερήσια ε, της ε, Ολομέλειας και έτσι να δείξουμε και στον κόσμο ότι προσπαθούμε να βελτιώσουμε πράγματα για την απάτη περί των ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο. Να δούμε αν θα γίνει οδηγία και κανονισμός. Στη, έχουμε στην σχετική οδηγία που υπάρχει τι θα γίνει με κάποιες ε, συναλλαγέ, ιδίως τις διασυνοριακέ, στα πλαίσια του προτινομένου κανονισμού Παίρνουμε ένα κεντρικό σύστημα ε, για πληροφόρηση για τις πληρωμές και έτσι να μπορούν τα κρατημέλη μελη να ξέρουν τι γίνεται με αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και αυτοί αλλά και τα κρατημέλη θα έχουν κάποιες υποχρεώσεις σε σχέση με αυτό το κεντρικό σύστημα διασταύρωση των πληροφοριών και έτσι να καταπολεμήσουμε την απάτη ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο είναι απαράδεκτο να υπάρχει απώλεια ε, εσόδων για τέτοιες συναλλαγές. Μιλάμε για πέντε δις ευρώ ετησίως. Δηλαδή, όλος ο τζίρο του ηλεκτρονικού εμπορίου της Πορτογαλίας το 18. 137 δις ευρώ το 2017 είχαμε πόλια εσόδων 266 ευρώ ανά Ευρωπαίο. Να, πώς έχει το σκηνικό. Άρα, θα πρέπει να βρούμε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα, σε αυτά τα προβλήματα και θα πρέπει να ληφθούν όλα αυτά υπόψη και από το Συμβούλιο ψηφιοποίηση γιατί εξελίσσεται η απάτη ε, και στα ψηφιακά τα πράγματα ε, δεν είναι, είναι πια πιο άειλα, πιο περίπλοκα και άρα θα πρέπει σιγά σιγά να έχουμε ένα τελείως ψηφιακό σύστημα ε, φορολόγησης οι φορολογικές αρχές να συνεργάζονται και πήγε ο διάλογος που υπάρχει να έχει αντίκρισμα, να ακολουθήσουμε τις καλύτερες πρακτικές, να συγχρονίσουμε τα συστήματά μας, τώρα όσον αφορά το, το blockchain και εδώ θα πρέπει να δούμε το θέμα της καινοτομίας, τώρα διακυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα βοηθήσει. Βελτιωμένη λειτουργία και το EDPS γιατί εδώ έχουμε όσον αφορά την προσθέτηση των δεδομένων κάποια δεδομένα που χρήζουν προστασίας. και χρειάζονται και εδώ υψηλά στάνταρ. Και τέλος αλλά σημαντικό, απλούστευση. Είναι ευκαιρία τώρα να απλουστεύσουμε κάποιες διαδικασίες. Πολύ σημαντικό για τον ΦΠΑ σε μια λογική ε, απλής προσωπικής υποβολής των δηλώσεων φόρου. Άρα, να αναδείξουμε τώρα το Κοινοβουλίο είναι πρόβλημα το πώς θα αλλάξει η Οικονομική Νομισματική Ένωση, να γίνει πραγματική ένωση, ένωση αγορών και αυτή η συζητούμενη πολιτική νοκρογωνίας λήθος φιλόδοξη να είναι η θέση του Κοινοβουλίου γιατί αυτό περιμένουν από εμάς οι πολίτες. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε, κύριο Μάρια Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την συνάδελφο για τη δουλειά που έκανε. Μια ισχυρή ευρωπαϊκή στρατηγική και διεθνή συνεργασία απαιτούνται για να πολεμήσουμε την απάτη του ΦΠΑ, όπου πολλοί παίζουν ένα σημαντικό ρόλο για να μειώσουμε το σχετικό κενό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο έκθεση σκοπεύει να βελτιωθεί η συνεργασία στην καταπολέμηση της σχετικής απάτης. Χαίρομαι για το ότι οι διάφορες ε, ιδέες ε, καλύπτονται ήδη και πλέον δεν χρειάζεται να υποβάλουμε τροπολογίες, οπότε εξ ονόματος των σοσιαλδημοκρατών μπορώ να πω ότι στηρίζουμε τις ε, τροπολογίες αυτές να κάνω δύο μόνο παρατηρήσεις. Όσον αφορά το πρώτο θέμα για τις απαιτήσει ε, για τους παρόχους υπηρεσιών, θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις γιατί αναβλήθηκε η ημερομηνία εφαρμογής ε, και σε σχέση με το άλλο θέμα για τα μέτρα που θα ενισχύσουν την διοικητική συνεργασία για να καταπολεμηθεί η φορολογική απάτη, θα πρότεινα να προσθεθεί μια αναφορά στην ε, οδηγία περί εξεπλήματος ε, χρήματος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ και εγώ. Κοβάρη από το Ρινιό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική του εργασία. Νομίζω ότι μπορούμε να στηρίξουμε πλήρως ε, την προσέγγιση της ε, σε αυτά τα δύο θέματα και να την ε, συγχαρούμε για τις προτάσεις της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο αναφέρθηκε στις σημειώσεις που διάσε ο μας ο κύριος Φέρμπερ είναι πάρα πολύ σημαντικό να φροντίσουμε η νομοθεσία μας να ταιριάζει με την ψηφιακή εποχή και βεβαίως ο εξυγχρονισμός που προσπαθούμε να κάνουμε να ταιριάζει με τις νέες τεχνολογίες αλλά και τους ε, νέους ε, τρόπους ε, απάτης. Οπότε αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς και πρέπει να φροντίσουμε να βρεθεί ο σχετικός τρόπος όσον αφορά τις υπηρεσίες τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ε, τεχνικές ε, παρατηρήσεις που νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντικές όταν μιλάμε για την εφαρμογή της νομοθεσίας και την αποδοχή από τους ενδιαφερόμενους. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι κανόνες που αφορούν τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών θα πρέπει να αφορούν μόνο τις πληρωμές στο διαδίκτυο γιατί αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος ε, διαφόρων κινδύνων ε, συμμόρφωσης. Επίσης σημαντικό είναι να φροντίσουμε να μην επιβάλλεται αχρίαστο βάρος στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών και επιπλέον να υπάρχουν τα σχετικά μέτρα που θα μας ε, βοηθήσουν να μην υπάρχουν διπλές αναφορές και τέλος καλό θα ήταν ε, να υπάρχουν αναφορές πιο συνολικές αντί ανά μία συναλλαγή ε, αρκεί βεβαίως να μην υπάρξουν παραθυράκια στην ε, νομοθεσία. Οπωσδήποτε θα δούμε τις δυνατότητες τροπολογιών προς αυτήν την κατεύθυνση και αναμένω την περαιτέρω συνεργασία με τον εισηγητή. Η κυρία Σκοτ πράσινη. Και εγώ θέλω πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω την κυρία Φερέρα για το σχέδιο εκθεσή τη ΣΥΜΕΣ και όδες εκ μέρους των Πρασινών. Όλοι ξέρουμε ότι οι απάτες που γίνονται για τι αγορέ. Ε, online είναι τεράστιες και οι απώλειες εκτιμώνται 5 δισεκατομμύρια το χρόνο από τις διασυνοριακές ε, τέτοιες συναλλαγές. Βέβαια, θα λειτουργήσει καλά το σύστημα εφόσον οι ενδιαφερόμενοι πληρώνουν τα τέλη και καταχωρούνται σε θελοντική βάση. Εμείς λοιπόν στηρίζουμε και είμαστε ευτυχείς με τις προτάσεις αυτές της Επιτροπής. Τώρα για τα όσα προτείνει η, η συγκήτρια. Δεν συμφωνούμε με τα τρία χρόνια, ούτε θέλουμε να υπάρξει αναβολή κατά δύο χρόνια για να αρχίσει να ισχύει η πρόταση αυτή. Η απάτη, όπως σας είπα, από το ΦΠΑ είναι τεράστια και πιστεύουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα όσο γίνεται πιο γρήγορα. Τώρα για τις δικές μας τροπολογίες. Μία πτυχή που μας απασχολεί είναι η δυνατότητα αξιολόγησης του αντικτυπού νέων νομοθετικών προτάσεων και κυρίως να δούμε πόσα χρήματα ε, εισπράχτηκαν τελικά ε, με τα νέα μέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελπίζουμε να έχει τα επόμενα χρόνια τις πληροφορίες που χρειάζεται για να μπορεί να υπολογίσει και τον αντίκτυπο αυτών των νομοθετικών προτάσεων. Ο κύριος Γιούσικα, PCR. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Εδώ είμαι. Η νομοθεσία για τα ΦΠΑ πρέπει όντως να αλλάξει για να καλυφθούν τα κενά. Οπότε χαίρομαι για τις προτάσεις. Όμως, έχω κάποιες επιφυλάξεις για την προτινόμενη νομοθεσία έτσι όπως την ανέφερε ο κύριος Σκοβάτσικ. Σύμφωνα με την Επιτροπή, τα κενά στο ΦΠΑ είναι της τάξης του 0,7% από αναμενόμενο ε, από τα αναμενόμενα έσοδα και σε μερικές χώρες φτάνει στα 35,5%. Πριν υπάρξει εναρμόνιση των κανόνων ΦΠΑ, θα άξιζε τον κόπο να αναλύσουμε και την αποτελεσματικότητα των εθνικών μέτρων καταπολέμησης της απάτης στο ΦΠΑ και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε γιατί μερικές χώρες έχουν τέτοιες διαφορές κατά 50 φορές μεγαλύτερες από όλες. Και τα μέτρα θα έπρεπε να είναι αναλογικά, χωρίς να επιβάλλουν επιπλέον διοικητικό βάρος στους παρόχους υπηρεσιών ε, πληρωμών. Τα ωφέλη από την νομοθεσία για την καταπολέμηση των απατών ΦΠΑ δεν θα πρέπει να είναι ε, υπερβολικά και να επιβάλλουν τεράστια γραφειοκρατία στις επιχειρήσεις. Φοβάμαι όμως ότι αυτό δεν ισχύει με την πρόταση αυτή που έχουμε μπροστά μας σήμερα. Η πρόταση λανθασμένα υποθέτει ότι εκείνος που πληρώνει έχει όλες τις λεπτομέρειες για τον τελικό δικαιούχο. Με κάρτες δεν γνωρίζουν οι τράπεζες απαραίτητα το IBAN. Οι μη ευρωπαϊκές χώρες δεν χρησιμοποιούν καθόλου IBAN Οπότε η πρόταση απαιτεί περισσότερες πληροφορίες από τους PSPs που ίσως δεν έχουν. υπερβολικό πάντως διοικητικό βάρος μπορεί να δημιουργήσει μειονέκτημα συγκριτικό και να επιβληθεί τελικά στους Ευρωπαίους καταναλωτές, χωρίς όμως να μειωθεί τελικά η απάτη θεωρώ πολύ σημαντικό ότι το αίτημα για πληροφορίες να περιλαμβάνει τις πληροφορίες εκείνες που εύκολα μπορούν να βρουν οι PSBs και να χρησιμοποιούνται για τη συλλογή δεδομένων όσον αφορά τον ΦΠΑ. Μία λύση για να μην υπάρχει τόση γραφειοκρατία ε, θα ήταν οι αναφορές κάθε συναλλαγής. Το μάλλον θα καταλήξει σε συμφωνία την Τετάρτη, έτσι κυκλοφορεί τουλάχιστον. Οπότε θα είναι μάλλον πολύ αργά για μας να επηρεάσουμε τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι επιφυλάξεις σχετικά με το κείμενο θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην θέση τη δικιά μας που θα πάει τελικά στο Συμβούλιο. Ευχαριστούμε. Σέτοβαν. Γκουε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο συνάδελφος ο κύριος Παπαδημούλης με παρακάλεσε να μεταφέρω τις ε, σκέψεις μας. Ε, πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε την εισηγήτρια για το σχέδιο έκθεσης μετά τον ε, κύριο Φέρμπερ που μετέφερε τις σκέψεις της και σας ευχαριστώ γι' αυτό συμφωνούμε όλοι ότι υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ πέρα με την απάτη του ΦΠΑ και επηρεάζονται τα κοινωνικά έσοδα και βεβαίως και οι φορολογούμενοι επιβαρύνονται αναλόγως. Οι αριθμοί που ανέφερε η Κομισιόν μιλάμε για 137 δισεκατομμύρια το 2017 Οπότε πρέπει να κάνουμε κάτι. Και δεν έχουμε κάνει αρκετά. Γιατί δεν υπάρχουν τα απαραίτητα πολιτικά μέσα ή δεν υπάρχει η απαραίτητη βούληση. Αλλά οπωσδήποτε χαιρόμαστε για το ότι οι περισσότεροι σκέφτονται κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση, ότι πρέπει δηλαδή να καταπολεμήσουμε την απάτη του ΦΠΑ με ενισχυμένη διοικητική συνεργασία, με ανταλλαγή δεδομένων, βέλτιστων πρακτικών, αλλά και την εισαγωγή νέων ε, τεχνολογιών. Και παρόλα αυτά, αυτά δεν επαρκούν για την ομάδα μας, δεν είναι αρκετά φιλόδοξα. Θεωρούμε ότι πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρές αποφάσεις από το Κοινοβούλιο να ενισχυθεί η διαφάνεια, η πρόσβαση στα δεδομένα, κάτι το οποίο βεβαίως ταυτόχρονα δεν θα πρέπει να αμφισβητεί τα προσωπικά δεδομένα. Εμείς θεωρούμε ότι επιχειρήσεις που έχουν ιστορικό τέτοια απάτης θα πρέπει να τιμωρηθούν και τέλος επιτρέψατε μου να πω εξ ονόματος του συναδέλφου Παπαδημούλη πως η κατανομή των αρμοδιοτήτων κάνει δύσκολο το να παίξει τον ρόλο του ως συνομοθέτη στο Κοινοβούλιο, στον τομέα της φορολογίας και πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά τα ζητήματα και έπρεπε να το έχουμε κάνει πιο νωρίς, όχι με αφορμή αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Οπότε... Δεν έχουμε αιτήματα για το KTI, οπότε δεν θα γίνουν κάποιες σχετικές ε, παρατηρήσεις. Ε, να σας υπενθυμίσω μόνο πως οι προθεσμοί για τροπολογίες είναι 11 Νοεμβρίου μέχρι τις 6 το απόγευμα. Η εξέτασή τους ε, θα είναι στις 2 Δεκεμβρίου και Δεκέμβριο επίσης θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Αυτό ισχύει και για τις δύο αυτές εκθέσεις. Οπότε περνάμε σημείο 9. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Πολ Τάγκ, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι η οδηγία αυτή τροποποιεί τις οδηγίες περί ΦΠΑ και ειδικών φόρων κατανάλωσης για να υπάρχει μια συνοχή στο πλαίσιο της ε, ΚΕΠΑ. Υπάρχουν ε, εξαιρέσεις ε, για τα κράτη-μέλη στον τομέα της ε, άμυνας μεταξύ όλων των κρατών μελών του ΝΑΤΟ. Με την δημιουργία της ΚΕΠΑ θα πρέπει βεβαίως να εξαιρεθούν και οι αποστολές ΚΕΠΑ από ΦΠΑ και ειδικού φόρους κατανάλωσης. και αυτό αφορά και το πολιτικό προσωπικό. Καθώς η οδηγία αυτή πλέον δεν επιτρέπει εξαιρέσεις και το ευρωπαϊκό δίκαιο απαγορεύει διαφορετική φορολογική μεταχείριση για διαφορετικούς δημόσιους φορείς που κάνουν το ίδιο καθήκον, είναι σημαντικό να το ρυθμίσουμε. Έκθεση λοιπόν της Κομισιόν απλά εισάγει την εξαίρεση της ε, ΚΕΠΑ ε, παράλληλα με αυτή του ΝΑΤΟ. Όσον αφορά την τεχνική φύση του κειμένου, το Συμβούλιο συμφώνησε γρήγορα σε μια κοινή θέση και δεν υπήρχαν σοβαρές ε, διαφωνίες όσον αφορά το περιεχόμενο αυτού του κειμένου. Οπότε προτείνω μια απλοποιημένη διαδικασία. Στην έκθεσή μου Έχω δύο ελάχιστες τροπολογίες. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά την διαβούλευση. για ζητήματα και παδεύτερον συμφωνώ με το Συμβούλιο για την θέση του εκτιμώντας 8 για την διευκρίνηση των πολιτικών μέτρων που δεν αφορούν άμεσα ζητήματα και ΕΠΑ τα οποία δεν πρέπει να επίπτουν σε αυτήν την εξαίρεση. Αυτά κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος κύριε Ντόρσαλ από το ΕΛΚ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστήσω τον συνάδελφο τον κύριο Τάγκ για την συνεργασία. Ε, ξεκάθαρη διαδικασία, τη στηρίζουμε. Έχουμε εδώ πέρα μια ευθυγράμμιση με αυτά τα οποία ισχύουν για το ΝΑΤΟ. Ε, πλέον ένα σημαντικό βήμα σε σχέση με την ΚΕΠΑ. Οπότε από εμάς πράσινο φως. Πρόεδρος. Κόβερικ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του και συμφωνώ ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η οδηγία για τους φόρους κατανάλωσης ε, για να ενημερωθεί όσο γίνεται και για την ε, ΚΕΠΑ σε σχέση με το ΝΑΤΟ. Θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με τις αμυντικές μας δυνατότητες. Θα πρέπει σε αυτόν τον τομέα να εξασφαλιστεί ότι υπάρχουν δίκαιοι όροι παιχνιδιού. Να μειώσουμε τη γραφειοκρατία, καθυστερήσεις φέρνει, είναι τροχοπέδι για τους στρατιωτικούς. Να κινηθούμε στα πλαίσια της ΚΕΠΑ και συμφωνούμε στο ότι θα πρέπει να υπάρξει ταχεία συμφωνία και να έχουμε την κοινή θέση του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε. Σκοτ Κέιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον Πολ Τάνκ, τον εισηγητή μας, γιατί έδειξε πνεύμα συνεργασίας. Συμφωνούμε. Απροστευμένη συνεργασία γιατί δεν υπάρχει κάτι επίμαχο η πράσινη θεωρούμε ότι σωστά να εξαιρέσουμε από τον ΦΠΑ τις κινήσεις της ΚΕΠΑ όπως και τις αποστολές του ΝΑΤΟ. Συμφωνούμε με τη σχετική τροπολογία στην ΣΕΝΤΕ. Να υπάρχει καταγραφή, παρακολούθηση, ακριβώς και οι επιχειρήσει ε, ωφελούνται τη απαλλαγή. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, γιατί όπως σας είπα, δεν υπάρχει κάποιο σημείο προστριβής. Ταχαίως να περάσει αυτό στο Συμβούλιο και να περάσει και στα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Γιούρζικα, του ECR. Θα είμαι σύντομος. Ευχαριστούμε και τον εισηγητή που ήταν πάρα πολύ γρήγορο στα όσα έκανε. Όπως είπαμε το Συμβουλίο ήδη έχει ε, συμφωνήσει και περιμένει να υπάρξει τελική ε, θέση. Ναι, να προχωρήσουμε με την απλουστευμένη διαδικασία γιατί είναι σημαντικό να ευθυγραμμίσουμε τις ε, ρυθμίσεις που υπάρχουν για τον ΦΠΑ, για τους έμεσους κατανάλωσης κλπ. Τι θα γίνει στην ΚΕΠΑ, τι θα γίνει στον ΝΑΤΟ, όλα αυτά όσο μπορούμε, όσο μπορούμε. Οπότε συμφωνούμε με την πρόταση του εισηγητού. Και είναι πάρα πολύ καλό το ότι υπάρχει μια ευρεία συνένεση για το θέμα της έκθεσης. Ο πρόεδρος, ευχαριστούμε. Σούντεβαν της Γκουα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον εισηγητή. Βεβαίω εμείς έχουμε διαφορετική πολιτική αξιολόγηση Βεβαίω έχουμε πιο επικριτική θέση ε, από όσα είπαν μέχρι τώρα οι συνάδελφοι για την ΚΕΠΑ και την οικοδόμηση μιας αμυντικής ένωσης. Εκτιμώ και την προσπάθεια του Πολτάγκ να υπάρχει σαφήνεια μεταξύ στρατιωτικών και πολιτικών αποστολών Παρ' όλα αυτά, σε γενικές γραμμές δεν ε, συμφωνούμε και άρα δεν συμφωνούμε με το να δούμε το θέμα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 52 σε επιταχυμένη διαδικασία. Εμείς θα υποβάλουμε τροπολογίες. Ευχαριστώ. Έχει προταθεί για την απλοποιημένη διαδικασία η έκθεση και αν δεν υπάρχει αντίρρηση από έξι μέλη της Επιτροπής μας για να χρησιμοποιηθεί η απλοποιημένη διαδικασία θα ισχύσει αυτή. Υπάρχει αντίρρηση. Θέλω να παρακαλέσω όσους ε, διαφωνούν ε, να σηκώσουν το χέρι. Οπότε δεν έχουμε φτάσει το όριο. Οπότε θα προχωρήσουμε με την απλοποιημένη διαδικασία όπως προτείνεται. Και η προθεσμία είναι Παρασκευή 15 Νοεμβρίου για οποιαδήποτε αντίρρηση. Συνεχίζουμε και πηγαίνουμε στο σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ετήσια έκθεση 2018. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μαυρίδη ε, από τους Σοσιαλδημοκράτες. Ο κύριος Μαυρίδης δεν είναι εδώ όμως. Οπότε σταματάμε για λίγο και θα επανέλθουμε σε τέσσερα λεπτά. So let's get started. Ωραία. Να αρχίσουμε λοιπόν με το σημείο 10 στην ημερήσια διάταξη. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Μαυρίδη, από τους σοσιαλδημοκράτες. Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μόλις έφτασα με το αεροπλάνο, ξέρετε από την Κύπρο δεν είναι εύκολο να φτάσει κανείς. Δεν υπάρχει απευθεία πτήση. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Έκθεση για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ετήσια έκθεση 2018. Η έκθεση αυτή αντικατοπτρίζει τις καλέ σχέσει που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι το κύριο μέσο που έχουμε για να εκφράζουμε τις απόψεις μας, αλλά και επικοδομητική κριτική σχετικά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη σταθερότητα τιμών, προκειμένου να υπάρξει πραγματική σύγκληση. Έτσι λοιπόν ετοίμασα και το σχέδιο έκθεσης για φέτος. Ο χρόνος έχει μεγάλη σημασία γιατί είναι η πρώτη τέτοια έκθεση για τη νέα αυτή θητεία και είναι και μετά την εκλογή τη νέα Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πρέπει λοιπόν να είναι ισορροπημένο το κείμενο, αλλά και χρήσιμο, επικεντρώνοντα στα εξή. Πρώτον, τι νομισματικέ αποφάσει τη ΕΚΤ το 2018 και τι επιπτώσει που είχαν στι οικονομίε τη Ευρωζώνη, όπω επίση και άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τι πολιτικέ τη ΕΚΤ και τι πρέπει να γίνει στη συνέχεια, όπω επίση και για τη λογοδοσία. Πιο συγκεκριμένα τώρα, για τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ του 2018 και τον αντίκτυπό τους στις οικονομίες Ευρωζώνης, ε, Ευχαριστούμε για τον ρόλο που έπαιξε η ΕΚΤ στη σταθερότητα και υπογραμμίζουμε ότι το πρόγραμμα αγοράς ε, ομολόγων έχει συνεισφέρει πολύ σημαντικά στην οικονομική ανάκαμψη. Επίσης σημειώνουμε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις επί των ε, τραπεζών έχουν αντισταθμιστεί προς το παρόν από τα ωφέλη μεγαλύτερου δανεισμού σε χαμηλότερο κόστος. Συγχρόνως υπογραμμίζουμε ότι είχαμε πολύ χαμηλά επιτόκια, πολύ κοντά στο μηδέν και αρνητικά που δίνουν ευκαιρίες στους καταναλωτές και τους ε, δανειζόμενους σε αυτήν τη δύσκολη στιγμή με χαμηλή απασχόληση και συγχρόνως εκφράζουμε την ανησυχία μας ότι μετά από μία σύντομη ανακαμψή έχει μειωθεί πολύ στο 1,2% του ΑΕΠ η αύξηση της ε, ανάπτυξης. Και συνεπώς τονίζουμε ότι πρέπει η νομισματική πολιτική να παραμείνει διευκολυντική για το προβλεπόμενο μέλλον. Κάτι άλλο σημαντικό που θέτει η έκθεση αυτή είναι σχετικά με το σύστημα κεντρικών τραπεζών και τους εμπειρογνώμονες οι οποίοι αναλύουν τις διαφορές ανάμεσα στην ανάκαμψη της αγοράς εργασίας και τους μισθούς οι οποίοι παραμένουν χαμηλοί. 6,2% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 7,4% στην Ευρωζώνη ήταν η αύξηση, το χαμηλότερο από το 2008. Αλλά αυτή η μείωση στην ε, απασχόληση δεν οδήγησε σε κάποια ανάπτυξη. Έπειτα έχουμε το Brexit, έχουμε την ε, Κεφαλαϊκή Ένωση, έχουμε τα κρυπτονομίσματα, τα πράσινα και άλλα ζητήματα. Από αυτά θα επικεντρωθώ σε δύο σημαντικά. Το πρώτο είναι η ολοκλήρωση της ε, Τραπεζικής Ένωσης με την αμεδιοποίηση του προγράμματος εγγύσεων και το δεύτερο έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή και τη Συμφωνία των Παρισίων, βάσει της οποίας δεσμεύεται η Ευρώπη και πρέπει να σέβεται την εντολή της και την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε σχέση με αυτά. Τώρα, για το μέλλον. Εμείς τονίζουμε ε, τις φορολογικές πολιτικές, οι οποίες είναι, συγγνώμη, τη δημοσιονομική πολιτική, η οποία είναι αναγκαία για να ενισχύσει τη νομισματική πολιτική της ΕΚΤ. Επίσης λέμε ότι ενισχύοντας το ρόλο του ευρώ μπορούμε να πετύχουμε τη σωστή ισορροπία. Τέλος, όσον αφορά την λογοδοσία. Χαιρόμαστε για την ενίσχυση της λογοδοσίας υπό την Προεδρία του Μάριο Ντράκη, αλλά εκφράζουμε και την επιθυμία μας να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη λογοδοσία και διάλογος με τη νέα πρόεδρο. Επίσης τονίζουμε και το θέμα του ορισμού των μελών του Εκτελεστικού Συμβουλίου και ζητάμε να υπάρχει μια shortlist με ε, ισορροπία ανάμεσα στους άντρες και τις γυναίκες. Έπειτα θέλουμε feedback ένα τμήμα από την έκτη για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσον αφορά την ετήσια έκθεση για το 2017 και ζητούμε αυτή η λογοδοσία να συνεχιστεί και να συνεχίζεται η δημοσίευση γραπτού feedback πάνω στα ψηφίσματα και την ετήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ΕΚΤ. Προσβλέπω λοιπόν σε συζήτηση σήμερα αλλά και στο μέλλον και σε επικοδομητική συνεργασία με τους σκιώδεις συζητητές και τα κόμματα. Ευχαριστώ. Εμείς Ευχαριστούμε. κύριε Μεφρέν από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστούμε κύριε εισηγητή για την άριστη εισηγησή σας για το σχέδιο έκθεσης. Είναι μια στέρεα βάση για τις συζητήσεις που θα κάνουμε αυτές που θα γίνουν σε πνεύμα ανοιχτού διαλόγου και πνεύμα συνεργασίας. Υπενθυμίζω, είναι απαραίτητο να είναι ξεκαθρό στην έκθεση ότι οι τροπολογίες να αφορούν την εντολή της τράπεζας. Θα καταθέσω σχετικά τροπολογίες. Και σύντομα να πούμε τι γίνεται με τα βασικά. Όπως το είπατε, είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρχει ανεξαρτησία της τράπεζας, έτσι θα εκπληρώσει την αποστολή της όσον αφορά την σταθερότητα των τιμών, θωράκιση του διεθνούς ρόλου του ευρώ σε σχέση με τους κινδύνους από τα κρυπτονομίσματα, καλύτερη κατανόηση των αποφάσεων της τραπέζας από τους πολίτες και τέλος πόσο σημαντικό είναι να συνεχίζονται οι προσπάθειες της τράπεζας για την αντίσταση στους κινδύνους του Ιντερνετ, της κυβερνοαπειλές. βρια συνένεση και εδώ και στην Ολομέλεια. Μα είναι το πρώτο μας μήνυμα της Κριστιαν Λαγκάρντ ως ε, κοινοβουλίου. Άρα, θα πρέπει να ε, ληφθούν υπόψη οι συστάσεις για να υπάρχει ένας διάλογος πάγιος, συνεχής με την Επιτροπή. Ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ, Γαρικάνο, από τους φιλελεύθερους. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα ευχαριστίες προς ε, τον εισηγητή. Πολύ καλή η δουλειά του. Θα συνεργαστούμε και έχω σύντομες παρατήρησεις από πλευρά της Ναι, συμφωνούμε όσον αφορά τα όσα καλά κάνει η Κεντρική Τράπεζα για τα επιτόκια, για το γενικά πώς βοήθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση να βγει από την κρίση Επίσης, σύμφωνα μαζί του, για τις διαρθρωτικές αλλαγές στα θεσμικά της Ευρωζώνης. Αυτό χρειάζεται, χρειάζεται να μπουν και οι τελευταίες πινελιές. για εγγύηση καταθέσεων κλπ. Όσον αφορά την ρευστότητα και τα άλλα. Επίσης είναι σημαντικό να έχει πιο σημαντικό ρόλο η δημοσιονομική πολιτική όπως και η νομισματική πολιτική και γι' αυτό είναι θετικό ότι και ο Ντραγκή και η κυρία Λαγκάρντ το ετώνησαν. Κάτι να προσθέσω ε, ως ε, επικριτικό. Η Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να προσπαθήσει περισσότερο στο θέμα της επικοινωνίας. Είναι πραγματικό το πρόβλημα πώς προβάλλεται η νομισματική πολιτική, ιδίω στην Γερμανία. Υπάρχει νομισματικός λαϊκισμός. Οι αποφάσεις υφίστανται κριτική, επιθέσεις, χωρι να υπάρχει μια κριτική με Άρα, θα πρέπει η κοινωνική πολιτική να βελτιωθεί από πλευρά τη τράπεζα. Α μας προβληματίσει αυτό. Παρακαλώ και ο εισηγητή να το σκεφτεί. Γιατί ακριβώ, ιδίω όσον αφορά τι τελευταίε αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου, είδατε τι υποδοχή έγινε στα κράτη-μέλη. Κύριο Γιακελίνα. Πράσινη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και τον κύριο Μαυρίδη για την ε, έκθεση. Θα ε, επανέλθουμε. Συμφωνούμε. Βεβαίω, ω πράσινη μετά όσα είπατε για τη Συμφωνία των Παρισίων, για το ότι θα πρέπει και την Τράπεζα κάτι να κάνει σε σχέση με τι σχετικέ συστάσει. Επίσης, σύμφωνα με το είπατε για την ισότητα των δύο φίλων και το ότι η ισότητα θα πρέπει να διέπει ε, τους διορισμούς. Πάντως, εμείς θέλουμε να τονιστεί περισσότερο πόσο κάνατε εσείς το ότι θα βλέπει η τράπεζα λάβει υπόψη τις επιπτώσεις κάποιων μέτρων. Όπως και τονιστεί σε άλλες ε, εκθέσεις πτήσεις. Μεταξύ άλλων πάντως γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα και άλλες ε, συνέπειες οι ανισότητες. Αρνητικά επιτόκια, κόστος ε, του ενεργητικού, επιπτώσεις σε σχέση με τους επενδυτές και κίνδυνος μετακύλησης των συνεπειών των αρνητικών στους ε, καταναλωτές. Ε, για αυτό και εμείς λέμε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί το ποιες είναι οι μακροπρόθεσμες συνέπειες των μέτρων της ε, Κεντρικής Τράπεζας και όσον αφορά επίσης ε, τους διεθνείς διακανονισμούς. Θα πρέπει τα στοιχεία, τα κρυπτοστοιχεία του ενεργητικού να μελετηθούν από την Κεντρική Τράπεζα και τα κρυπτονομίσματα γιατί έτσι θα πρέπει να το βλέπουμε, όχι ως κρυπτονομίσματα, ως κρυπτοενεργητικό και θα κατεβάσω σχετική τροπολογία. Πέραν αυτό. Πρέπει η τράπεζα να προσπαθήσει μαζί με τις άλλες τράπεζες να δει τι ευκαιρίες, τι κίνδυνοι υπάρχουν σε σχέση με ψηφιακά νομίσματα, γιατί υπάρχουν εφαρμογές, ούτως ώστε να προστατευτεί περισσότερο ε, το τραπεζικό σύστημα. Στην έκθεση αναφέρει η τράπεζα και θα κάνω μια τροπολογία αυτό το καινούριο benchmark που αφορά τα προχειπρόθεσμα επιτόκια τελευταίο και σημαντικό. Συμφωνούμε. Θα πρέπει να κληρωθεί η τραπεζική αγορά, να επιταχύνουμε τις προσπαθίες μας τόσο να έχουμε περισσότερη χρηματοοικονομική ολοκλήρωση, να εκμεταλλευτούμε τα όσα έχουν προκύψει από λαθεσμικά όργανα ή από ακροάσεις. Καλά, μην κολλούμε στο θέμα της εντολής της ε, Κεντρικής Τράπεζας, το θέμα είναι ευρύτερο, αλλά θα πρέπει να έχουμε μια αρχιτεκτονική εποπτική πιο ομοιογενή. Είναι πολύ σημαντικό για τα χρηματοοικονομικά, για την ενιαία αγορά γενικότερα. Και πάλι συγχαρητήρια, θα συνεργαστούμε και να έρθουμε σε επαφή και με την τράπεζα για το μέλλον. Επόμενο. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω γερμανικά. Δεν θα σας προξενήσει η έκπληξη ότι δεν είμαστε πολύ θετικοί απέναντι σε αυτήν την ε, έκθεση. Δεν ανταποκρίνεται, θεωρούμε, στην εντολή της ε, ΕΚΤ. Ούτε είναι σωστή εκτίμηση όσον αφορά την επίδραση της πολιτικής της ΕΚΤ, αλλά δεν θέλω τώρα να μιλάω όλο το βράδυ, οπότε θα κάνω κάποιες λίγες σύντομες ε, παρατηρήσεις για τα σημεία στα οποία θα θέλαμε αλλαγέ. Πρώτον, πράσινα ομόλογα. Τα λεγόμενα αυτά ομόλογα τα φιλικά προς το κλίμα. Ε, λυπάται η έκθεση για το ότι μόλις 1% των ομολόγων σε ευρώ είναι πράσινα ομόλογα και αναφέρεται και στην έκθεση και στην Συμφωνία των Παρισίων. Όμως ε, η υποχρέωση που προκύπτει από την Συμφωνία των Παρισίων σαφώς δεν είναι αποστολή της έκτη αποστολή που καθορίζεται ξεκάθαρα στις συνθήκες στο άρθρο 127 μάλιστα για τη συνθήκη λειτουργία τη Ευρωπαϊκής Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει κατά κύριο λόγο να ασχολείται με τη σταθερότητα των τιμών. Και έχει και έναν δευτερεύοντα ρόλο στον συντονισμό της οικονομικής πολιτικής. Και τίποτα άλλο δεν είναι δουλειά της. Αυτά τα λένε οι συνθήκες. Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο τον σαφή ορισμό δηλαδή της εντολής της ΕΚΤ ε, απορούμε και για τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρονται που από ό,τι φαίνεται ε, είναι μια προσπάθεια να επεκταθεί η εντολή της ΕΚΤ με βάση πολιτικά κίνητρα. Τι εννοώ συγκεκριμένα. Πρώτα απ' όλα η δημοσιονομική ικανότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή αυτό το οποίο πιο είναι ε, πιο γνωστό ως ε, πρόταση για έναν προϋπολογισμό της Ευρωζώνης. Ούτε αυτό αναφέρεται πουθενά στις συνθήκες. Ε, δεύτερον, έχουμε σοβαρές επιφυλάξεις ε, όσον αφορά το έντις, ε, την δημιουργία δηλαδή μιας πανευρωπαϊκής ε, εγγύησης καταθέσεων και εξίσου επιφυλακτική και απορριπτική είμαστε όσον αφορά τις προσπάθειες δημιουργίας ευρωομολόγων υπό νέο όνομα. Και τέλος μια παρατήρηση από εμένα είναι αξιοσημείωτο σε ποιο βαθμό ακριβώς ε, τα αριστερά κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, ακολουθούν ε, την, και επενούν την πολιτική ενό ανθρώπου της Wall Street, του λεγόμενου Ντραγκιαβέλη, παρά το ότι αυτή ευνοεί τους πλουσιότερους στην κοινωνία και αργά αλλά σταθερά καταλήγει να στίβει την μεσαία τάξη. Και βεβαίω αυτά μας κάνουν να απορούμε και για το ΕΛΚ και τους επένους που προερχόνται από εκεί. Όπως σας είπα όμως δεν θέλω να μιλάω όλο το βράδυ, οπότε αυτά. Thank you. Ευχαριστούμε. Ο κύριο Σέπινγκ, ECR. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω Ολλανδικά. Γιατί διαβάζω εδώ εκ μέρου του κύριου Φανόφαλτβεντ, που είναι σκιώδη εισηγητή. Ο σκιώδη εισηγητή, ε, λοιπόν, δυστυχώ δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα γιατί είναι σε τριμερή διάλογο όσον αφορά τον προπολογισμό του 2020 και επειδή είναι πρόεδρος στην Επιτροπή Προπολογισμών έπρεπε να είναι εκεί. Ο κύριος Φανόφερφελτ λοιπόν μου ζήτησε να τον συγχωρήσουμε που δεν είναι εδώ. Μου έδωσε κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά την έκθεση του κύριου Μαυρίδη. Και θα σας πω ποια είναι αυτά τα σημεία. Πρώτον, όσον αφορά την ανεξαρτησία τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ο κ. Φανόβερο Φέλτε λέει ότι πράγματι έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και δεν πρέπει να πολιτικοποιηθεί το όργανο και να επηρεάζεται από την πολιτική. Δεύτερον, λέει ότι η πολιτική προϋπολογισμού επηρεάζεται από την νομισματική πολιτική θα πρέπει να υπάρχει κάποια αντιστάθμιση ανάμεσα στην νομισματική και τη δημοσιονομική πολιτική, πότε είναι επεκτατική μία ή άλλη. Και σε περιπτώσεις κρίσης θα πρέπει μία να ενισχύει την άλλη. Για να μην είμαστε σε μία κατάσταση που να απαιτείται σύγκληση των δύο. Επίσης, μιλάει για την ομάδα εμπειρογνωμόνων όσον αφορά την απασχόληση, ότι χρειάζεται καινοτομία και ευελιξία για να είναι ανταγωνιστική. Δεν θα πρέπει να θεωρούνται αρνητικές τέτοιες εξελίξεις. Χρειάζεται επίσης αύξηση της παραγωγικότητας, και να ξέρουμε ότι μόνο όταν υπάρχουν χαμηλότερη η μισθή μπορεί να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα. Επίσης, όσον αφορά την, την ε, Τραπεζική Ένωση, πιστεύει ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρωθεί. Και το σύστημα εγγύσεων πρέπει να γίνει πραγματικότητα, αλλά μόνο όταν έχουμε προχωρήσει περισσότερο και έχουν μειωθεί δραστικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πέμπτον, ο κύριος Φανόφερβελτ Όσον αφορά την νομισματική πολιτική, πιστεύει ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες επικρίσεις. Ότι τα αρνητικά αποτελέσματα ή τα περιορισμένα και ότι όσον αφορά τις ευκαιρίες που έχουμε χάσει, όντως η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει χάσει κάποιες ευκαιρίες ότι μπορούν να υπάρξουν στο μέλλον παρετέρω τροποποίησης Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σίδεβαν της ΓΚΟΕ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αντικαθιστώ τον κύριο Παπαδημούλη εδώ με παρακάλεσε να μεταφέρω τις ε, σκέψεις του. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον κύριο Μαυρίδη για το σχέδιο έκθεσης ε, το οποίο περιέχει στοιχεία με τα οποία μπορούμε να συμφωνήσουμε. Μου ζήτησε όμως ο κύριος Παπαδημούρης να κάνω κάποιες ακόμα παρατηρήσεις ε, που θεωρούμε απαραίτητες Πρώτα απ' όλα πρέπει να τονιστεί ότι χρειαζόμαστε ανάπτυξη και πρέπει να ξεπεραστούν τα κένα που υπάρχουν στις περιφέρειες, στις επενδύσεις Γι' αυτό θα πρέπει να αυξηθούν οι δημόσιες επενδύσεις και ταυτόχρονα να δούμε την περιφερειακή και κοινωνική συνοχή και την ποιοτική απασχόληση με καλές δουλειές. Και βεβαίως αυτό πάντα με την βοήθεια της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής ε, Τράπεζας. Ε, επίσης ο κύριος Παπαδημούλης μου ζήτησε να υπενθυμίσω ότι πρέπει να επιμείνουμε στην εκμετάλλευση όλων των δυνατοτήτων που μας δίνει το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, αλλά για εμάς είναι απολύτως απαραίτητο το σύμφωνο αυτό να συμπληρωθεί, να αντικατασταθεί στο προσεχές μέλλον από ένα σύμφωνο ανάπτυξης και απασχόλησης. Επίσης θα πρέπει να δοθεί περισσότερο βάρος στην ενισχυμένη διαφάνεια, δημοκρατική λογοδοσία και πάντα τηρώντας την ανεξαρτησία της ΕΚΤ. Και βεβαίως ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει οι συστάσεις ε, της Ευρωπαίας ε, Διαμεσολαβητού να ληφθούν υπόψη ε, από τον κύριο Ντράγκη και την ε, διαδοχό του. Βλέπουμε πως υπήρχαν κάποιες αξιολογήσεις και χαιρόμαστε για την ξεκάθαρη τοποθέτηση της ΕΚΤ και του εισηγητή εδώ πέρα για μια ευρωπαϊκή εγγύηση καταθέσεων για να προστατεύσουμε τους αποταμιευτές και θετικό είναι το ότι η κυρία Λαγκάρτ υποσχέθηκε να συνεισφέρει θετικά στην προστασία του κλίματος. Οπότε σας ευχαριστούμε για όλα αυτά και θα υποβάλουμε τις τροπολογίες μας στις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Κύριε Μαυρίδη, θέλετε να κάνετε κάποιες τελικές listened. Απλώς να πω ότι άκουσα μεγάλη προσοχή και περιμένω τι ε, τροπολογίε και τη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Okay, so... Πρόεδρος, καλώς, οπότε για τι τροπολογίε έχουμε την 12η Νοεμβρίου το μεσημέρι ως καταληκτική ημερομηνία και προθεσμία για τις τροπολογίε και Έχουμε ανοιχτή ε, συνεδρίαση για τους συντονιστές με συμμετοχή της κοινή αντιπροσωπείας στις 6.30 στο PHS 6Β54. Ανοιχτή συνεδρίαση για όλους τους συναδέλφου το προσωπικό και επόμενη συνεδρίαση Έκον Λίμπε, κοινή συνεδρίαση 5η στις 7 Νοεμβρίου. 11.30 με 12.30 για καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος και επόμενη συνεδρίασή μας Δευτέρα 18 Νοεμβρίου στις 3 το απόγευμα. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.